Minister, thank you very much for coming. This is time to make an assessment of your presidency of the Council of the Union. We have uh, with us... Uh, Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νεοκλή Σιλικιώτη, ο οποίος είναι υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ομιλία του μεταδίδεται στο διαδίκτυο σε ένα ευρύτατο ακροατήριο εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας. Θα μας μιλήσει λοιπόν στον τομέα της πολιτικής διεθνούς εμπορίου. Ε, η Κυπριακή Προεδρία ήταν πάρα πολύ δραστήρια στον τομέα του εμπορίου και επέτυχε να ολοκληρώσει ορισμένους πολύ ευαίσθητους φακέλους αρχίζοντας με το εξαιρετικό φάκελο της ε, συνεργασίας με το Πακιστάν επίσης ε, την ε, διμερή ρήτρα διασφάλισης και τη μηχανισμό σταθεροποίηση με την Κολομβία και το Περού, τη συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά το πακέτο Omnibus, το οποίο πριν από την Κυπριακή Προεδρία ήταν κατά κάποιο τρόπο παγωμένο. Είχε παγώσει. και υπό την Κυπριακή Προεδρία αναζωογονήθηκε και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας που ξεπαγώσατε αυτό το φάκελο. Ήμουνα ένα ήταν ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία είπα στον Υπουργό κύριο Σικλιώτη και είχα πει ότι ανησυχούσα ιδιαίτερα για την εξέλιξη του φακέλου Omnibus και ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω ότι πραγματικά θα υπάρξει μια πολύ σημαντική πρόοδος σε αυτούς τους φακέλους. Είναι ένα ορόσημο θα έλεγα αυτή η πρόοδος και ένα ορόσημο της προηδίας σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και έχετε άνεση χρόνου να παρουσιάσετε την ε, ομιλία σας και επίσης για τη συζήτηση. Ευχαριστώ ε, Ευχαριστώ κύριε Θα μιλήσω στα ελληνικά. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, όταν τον περασμένο Ιούλιο αναλάβαμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας παρουσίασα τις βασικές μας προτεραιότητες και τα θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε, όπως αυτά είχαν καθοριστεί μέσα στο πλαίσιο του τρίου της Προεδρίας, Πολωνία, Δανία, Κύπρος. Σήμερα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εξάμεινη θητεία της Κυπριακής Προεδρίας, επανέρχομαι για να σας παρουσιάσω τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Η σημερινή συνοπτική παρουσίαση του έργου που επιτελέσαμε κατά τη διάρκεια της εξάμενη ιδίας μας έχει συνεπώς μια διάσταση λογοδοσίας της Προεδρίας του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα όμως εξυπηρετεί και μια αναγκαινότητα, ότι δηλαδή στη δράση και στις πολιτικές που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης αλλά και η εναλλακτική μορφή ισχύω που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνέ σκηνικό έχουν ω αφετηρία μια κίνηση συνισταμένη. Αναγάγαμε το διεθνέ εμπόριο ω την αιχμή του δόρατο, αλλά και ω ισχυρό μοχλό τόσο για την εδραίωση δικαιότερων κανόνων στο παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό σύστημα, όσο και για την πρόθεση και υπεράσπιση θεμελιώδων αρχών και αξίων, όπως είναι η δημοκρατία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει φέρει αντιμέτωπη την Ευρώπη με σημαντικές προκλήσεις και άμεσες αρνητικές επιδράσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει και να διατηρήσει το χαρακτήρα και την ταυτότητά της ως μια οντότητα που παραμένει αλληλέγγυα προς τα κράτη και τους λαούς. Για αυτήν την καλύτερη Ευρώπη η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε έντιμα, με συνέπεια και ακούραστα τους τελευταίους έξι μήνες και σε αυτήν την Ευρώπη θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία να ανήκει και να υπερασπίζεται. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το οικονομικό σκηνικό στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δυσμενές. Η εξέβρεση τρόπων αντιμετώπισης κρίση συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, η πεποίθησή μας ήταν και θα παραμένει ακλόνητη για τη συνεισφορά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το διεθνές εμπόριο για αντιστροφή αυτής της κατάστασης. Όπως σας είχα αναφέρει και στην αρχική μου παρέμβαση τον Ιούλιο, το διεθνές εμπόριο αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για την ανάκαψη και την αθέρμανση της οικονομίας. Θα ήθελα μάλιστα να επαναληφθήσω αυτή τη σημασία επικαλούμενο τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, του κ. Πασκάλ Λάμι, ο οποίο στην πρόσφατα δημοσιευθήσα ετήσια έκθεση του οργανισμού είπε ότι χρειάζεται μια ανανεωμένη και ισχυρότερη δέσμευση από όλες τις κυβερνήσεις για να αναζωογονηθεί το πολυμερές εμπορικό σύστημα και να αποκατασταθεί η οικονομική ασφάλεια σε μια χρονική στιγμή που είναι απολύτως αναγκαία. Συνειδητοποιούμε αυτή την πραγματικότητα, συνειδητοποιούμε δηλαδή το γεγονό ότι ακόμα και η παραμικρή εξέλιξη στον πόριο μπορεί να τονίσει την ανάπτυξη και κατ' επέκταση να ενισχύσει την οικονομία μα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια τη Κυπριακή Προεδρία, προσπαθήσαμε να δώσουμε όθηση και να προωθήσουμε τα θέματα διεθνούς εμπορίου, ώστε απρόσκοπτα να προάγεται η ανάπτυξη του εμπορίου τόσο με στρατηγικούς εμπορικούς μας εταίρους, όσο και με άλλες σημαντικές οικονομίες. Πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη, με τη σκληρή μας δουλειά και τη στενή συνεργασία που είχαμε με όλα τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει και να συμβάλλουμε στην επιτυχή πρόοδο σημαντικού αριθμού εμπορικών θεμάτων. Θα ήθελα πρωτού προχωρήσω να εκφράσω την εκτίμηση και τις θερμέ μου ευχαριστίε προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα προς εσά, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνού Εμπορίου, αλλά και σε εσά προσωπικά, καθηγητή Μορέιρα, για την επικοδομητική συνεργασία και σημαντική συμβολή που είχατε για την επιτυχή κατάληξη πολλών φακέλων που διαχειριστήκαμε αυτή την περίοδο. Θα αρχίσω τον απολογισμό αναφερόμενο στου νομοθετικού φακέλου, για την πρόθεση των οποίων από την αρχή είχαμε θέσει ω βασικό στόχο την ανάπτυξη ουσιαστική και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θεωρώ ότι έχει διαφανεί από τι πρώτε μέρε ανάληψη τη Προεδρία μα, όταν ανταποκριθήκαμε άμεσα στι ανησυχίε του Κοινοβουλίου όσον αφορά εκτελεστικέ διατάξει που περιλαμβανόταν σε αποφάσει του Συμβουλίου για ολοκλήρωση διεθνών συμφωνιών, οι οποίε έπρεπε να υιοθετηθούν με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η αποτελεσματική επίλυση του θέματος αυτού επέτρεψε την εξασφάλιση χωρίς καθυστερήσει της συνέδεση του Κοινοβουλίου για την εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, τη συμφωνία σύνδεση με τις χώρες της Κεντρική Αμερικής, τη συμφωνία για εξαγωγές ξυλίας από τη Ρωσική Νομοσπονδία καθώς και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ σχετικά με την αξιολόγηση συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλα, μέσα σε πνεύμα συνεργασία και συνένεση με το Ευρωκοινοβούλιο, έχει επιτευχθεί συμφωνία σε σημαντικού νομοθετικού φακέλους όπως οι κανονισμοί για την εφαρμογή διμερούς ρήτρα διασφάλιση του μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε στο πλαίσιο τη εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και τον Περού και τη συμφωνία σύνδεση με την Κεντρική Αμερική. Ο κανονισμό για τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στι εξαγωγέ ξυλία από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η τροποποίηση του βασικού κανονισμού αντιτάπινγκ. Ο κανονισμό σχετικά με την τροποίηση και συμπλήρωση του παρακτήματο 1 του κανονισμού 2658 κάθετο 87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Και τέλο και φυσικά ο κανονισμό για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτη ανάγκη στο Πακιστάν, για τον οποίο ομολογουμένω αρκετή πρόοδο έχει επιτευχθεί κατά την προηγούμενη Διδανική Προεδρία. Επιπρόσθετα, έχουμε εργαστεί σκληρά προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στι προτάσει κανονισμών Omnibus 1 και Omnibus 2 σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για εμπορικά θέματα στι προνοιε τη συνθήκη τη Λισαβόνα όπως είχαμε δεσμευτεί βεβαίω από την αρχή και είμαι ευτυχή γιατί κατά την Προεδρία μα έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση κοινή θέση του Συμβουλίου για την πρόταση κανονισμού Omnibus 1 και έχουν ήδη ξεκινήσει οι τρίλογοι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά στο Omnibus 2, είμαι πεμπισμένο ότι με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το Συμβούλιο θα μπορέσει πολύ σύντομα να διαμορφώσει τη θέση του και να ξεκινήσει τριλόγου με το Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια τη Κυπριακή Προεδρία έχει κατά την άποψή μου επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος και στις διαδικασίε σύναψης διμερών εμπορικών συμφωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ως σημαντική επιτυχία θεωρείται η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου στις 29 Νοεμβρίου των διαπραγματευτικών εντολών για σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Η ελόγω συμφωνία είναι τεράστια σημασία για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού βάσει εκτιμήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ένωσης κατά περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχοντας επίγνωση ότι το θέμα των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τα κράτη-μέλη, ως Προεδρία προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ενεργώντας ως έντιμοι μεσολαβητέ, το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα που να διασφαλίζει τα συμφέροντα των κρατών μελών αλλά και να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε διασφαλίσει την τήρηση των αναγκαίων ισορροπιών στις διαπραγματευτικές εντολές ώστε να προφυλάσσεται τόσο η βιωσιμότητα των εξαγωγικών αγορών της Ευρώπης ως σύνολο όσο και τα εμπορικά συμφέροντα σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομεί των κρατών μελών. Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι στις διαπραγματευτικές εντολές που το Συμβούλιο έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και οι δικές σας θέσεις όπως περιέχονται στο σχετικό για το θέμα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Μια από τις οριζόντιες προτεραιότητες που είχε θέσει η Κυπριακή Προεδρία ήταν η δυνάμωση και ανάδειξη της μεσογειακής διάστασης των πολιτικών έτσι, στο πλαίσιο τη ευρωμεσογειακής συνεργασία δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τι χώρε τη νότια Μεσογείου. Η απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη σφαιρική και σε βάθο συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Μαρόκο είναι το πιστέγασμα των προσπαθειών τη Κυπριακή Προεδρία. Αναμένουμε επίση ότι στου επόμενου μήνε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίε που βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να ξεκινήσουν σύντομα και οι διαπραγματεύσεις με την Τινησία. Όσον αφορά στι ε, εξελίξει διαπραγματεύσει για περιεκτική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, απομένει πολύ μικρό αριθμός εκκρεμούν των θεμάτων και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα οι διαπραγματεύσει θα ολοκληρωθούν. Είναι ίσω περιττό να αναφέρω ότι η ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων θα μας αποφέρει μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εύστοχα έχει λεχθεί, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίω. Παράλληλα, μια επιτυχή συμφωνία θα στείλει έναν ισχυρό μήνυμα για τη συνεχή προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ανοιχτές αγορές όσο και στο διατλαντικό χώρο και θα αποτελέσει πολύτιμο σημείο αναφοράς στις μελλοντικές μας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Χαιρετίζουμε επίσης την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με τη Σιγκαπούρη, των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα στείλει ισχυρό μήνυμα σχετικά με, τις, με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία με την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού και θα επιβιώσει την προσήλωσή της για εμβάθυνση των εμπορικών της σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρω διαπραγματεύσεων με το Βιετνάμ. Στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης έχουν προχωρήσει σημαντικά οι διαπραγματεύσεις για σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με την Αρμενία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία και ευελπιστούμε σε ολοκλήρωσή του τον κατάλληλο χρόνο. Αναφορικά με τις υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ιδία, καταβλήθηκε από πλευρά μα κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδο. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, αναγνωρίζουμε ότι ενδεχόμενη συμφωνία παρουσιάζει σημαντικέ ευκαιρίε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι διαπραγματεύσει οδηγήσουν σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Στα πλαίσια των διμερών σχέσεων έχουμε ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε ό,τι αφορά στην τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών αμοιβίας αναγνώριση σε σχέση με την αξιολόγηση πιστότητα, τα πιστοποιητικά και τη σήμαση πιστότητα. Κυρίε και κύριοι, η ανάπτυξη και φιλελευθερωποίηση του εμπορίου με στρατηγικού μα εταίρου και η καλλιέργεια στενέτερων σχέσεων έχει τεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα τη Προεδρία μα. Η ΕΠΑ αποτελούν το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε εμβάθυνση της συνεργασίας μας ε, μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφέλη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της απασχόλησης και ανάπτυξης μελετάται από την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου και αναμένεται η τελική έκθεση εντός των επόμενων εβδομάδων. Βάσει των προκαταστικών προτάσεων τη ομάδα εργασία αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για σύναψη συμφωνία ελευθέρων πορεία με τι ΗΠΑ εντό του επόμενου έτου. Όσον αφορά στην Κίνα, με την οποία οι εμπορικέ προοπτικέ είναι σαφώ μεγάλε, μετά από τη συζήτηση που είχαμε στη διάρκεια του γεύματο στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σχηματισμό Υπουργών Εμπορίου, διαφαίνεται ότι υπάρχει και το κατάλληλο κλίμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη για διερεύνηση της έναξης διαπραγματεύσεων επενδυτικής συμφωνίας. Στη συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνεται και η πρόσβαση στην αγορά αφήνοντας σε μετέπειτα στάδιο οποιαδήποτε συζήτηση για συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, κάτι το οποίο έχει προταθεί από την κινέζικη πλευρά. Σχετικά με τη Ρωσία, κατά διάρκεια της Προεδρίας μας δόθηκε έφαση στην αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία και στην εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ρωσίας μετά την προσχώρησή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τα θέματα αυτά μας, μας απασχόλησαν επίσης και κατά τη συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου τον περασμένο μήνα. Η γενική αντίληψη που επικράτησε ήταν ότι οποιασδήποτε παρεκκλήσεις της Ρωσίας από τις πολυμερείς αλλά και διμερείς δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, κατά την άλυψη της Προεδρίας μας, ήταν ήδη γνωστό ότι οι διαπραγματεύσει σε πολυμερές επίπεδο βρίσκονται σε μια διάμεση φάση. Κατά συνέπεια, σε αυτού του έξι μήνε οι προσπάθειέ μα επικεντρώθηκαν στη δημιουργία συνθηκών που θα δώσουν νέα δυναμική στο γύρο τη Στόχα με την πρόθεση των διαπραγματεύσεων στου λεγόμενου τομεί πρώιμης συγκομιδής, όπως η διευκόλυνση εμπορίου, η συμμετοχή των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, καθώς και μια πλειονομερή συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας έχουν ληφθεί ουσιαστικές αποφάσεις που αφορούν στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα αναφέρω ενδεικτικά τις αποφάσεις για ένταξη του Λάους και του Τατσικιστάν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα για τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ΚΑΤ στο πλαίσιο της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη σύναψη συμφωνιών με τη Βραζιλία και Ταϊλάνδη για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη Ευρωβουλευτέ τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έχω ήδη αναφέρει και στην αρχή, εργάστηκε για μια καλύτερη Ευρώπη. Αυτό αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα των προσπαθειών μα σε όλου του τομεί. Στο διεθνέ εμπόριο, το τελευταίο εξάμεινο λήφθηκαν σημαντικέ αποφάσει και έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδο σε μεγάλο αριθμό θεμάτων, ενώ έγινε κατορθωτή η επίτευξη συμφωνία σε κρίσιμου φακέλου. Αυτό το γεγονό μα επιτρέπει να αισθανόμαστε ότι παρά το μικρό μα μέγεθο ω χώρα, έχουμε συμβάλει στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και προποθέσεων για τόνωση τη ανάπτυξη και την ανάκαμψη τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγμα με τη σκητάλη, νιώθοντα ικανοποίηση για τα όσα έχουν επιτευχθεί για τον κοινό ευρωπαϊκό καλό με γνώμονα πρώτα και κύρια τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχόμαστε σύντομα να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο κοινή ιστορίας που να καταγράφει άρθηση, ευημερία και ανάπτυξη όπως ακριβώς το συνέλαβα οι οραματιστές του Ευρωπαϊκού Αυτού Δεν έχω παρά να ευχηθώ στο επόμενο τρίο της Προεδρίας και ιδιαίτερα στην Ιρλανδία ως η επερχόμενη χώρα κάθε επιτυχία. Ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μορέιρα και τα μέλη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τη συνεργασία, να ευχαριστήσω από αυτά τα μέλη τον Επίτροπο Αντιακού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθεια της, όλα τα κράτη-μέλη που συνέβαλα στο να έχουμε ολοκληρώσει αυτόν το εξάμεινο την Προεδρία μας, αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από αυτόν το βήμα τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εμπορίου Μηχανές και Τουρισμού, που συνέβαλαν τεμέγιστα μέσα από τη δουλειά του στι ομάδε εργασία, του λειτουργού των Χαράλαμπων Ρούσων, τον Χρήστο Παντελή και τον Γιώργο Τσαμέτη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Minister, for your comprehensive expose of uh, your six months in εξαμήνου της Προεδρίας σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Το πρώτο αίτημα από την κυρία Γκέλερ, τον Πρασίνα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μας παρουσιάσατε τις, ε, τα επιτεύγματα της Κυπριακής ε, Προεδρίας σε πολύ ενδιαφέροντους καιρούς. Έχω κάποια ερωτήματα στις διάφορες συμπορικές συμφωνίες που αναφέρατε. Και θα ήμουν γνώμη αν μπορούσατε να μας πρόσετε τις ιδέες σας. Καθαρά, σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Η συμφωνία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό που απομένει να επιληθεί είναι το ζήτημα της διασύνδεσης του Καναδά με την άμεση πρόσβαση σε ό,τι αφορά το βόλιο και χείριο κρέας σε σχέση με το συνολικό ε, κεφάλαιο των ηλεκτρονικών προμηθειών ε, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε το, το καναδικό αίτημα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα ήταν να περάσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές που έχει θέσει το Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε πώς συζητείτε αυτό στο Συμβούλιο και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Και μήπως επίσης θα μπορούσατε να μας εγγυηθείτε ως Κυπριακή Προεδρία, εξ ονόματος δηλαδή του Συμβουλίου, πρώτα απ' σε περίπτωση ότι δοθεί ελεύθερη πρόσβαση του βόηου και χείριου κρέατος θα έρχεται στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη ε, σεβασμό των ε, συνθήκων σε ό,τι αφορά τις τις ε, συνθήκες και τους όρους ε, ασφαλείας ε, που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που αφορούν τη συνθήκη και τη συμφωνία σε ό,τι αφορά τα θέματα πνευματικής διοκτησίας θα γίνουν επίσης σεβαστές οι σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το επόμενο θέμα σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί σχετικά, αλλά ακούσαμε ότι το Συμβούλιο άλλαξε την προκαταρτική εντολή που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον όντω συμβαίνει και κατά ποιον τρόπο έχει αλλάξει το προσχέδιο αυτό της εντολής και ιδιαίτερα το κατά πόσον έχουν τεθεί επιπρόσθετοι όροι σε ό,τι αφορά την Ινδία, αναφέρατε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος. Μπορείτε να εξηγήσετε ποια υπήρξε αυτή η πρόοδος, γιατί νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο ε, στάση αυτή τη στιγμή. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τη Σιγκαπούρη, επίσης αναφέρατε ότι τον Φεβρουάριο δεν δόθηκε καμία λύση σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό εφαρμογής, το πώς θα εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών στην ε, ε, παρακολούθηση εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας. Έχουν επιληθεί τα ζητήματα αυτά και είστε θετικοί σε ό,τι αφορά την συμφωνία αυτή και με δεδομένη τη δυσκαλία της ε, κυβέρνησης της, ε, ε, της κυβέρνησης να αποδεχθεί την ελεύθερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον ο μηχανισμός εφαρμογής και παρακολούθησης συμφωνίας είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Ευχαριστούμε. Πολύ καλά ερωτήματα. Άλλα. Από, τα... από το κρατήριο. Εγώ έχω να υποβάλω μια σειρά ερωτημάτων. Σε ό,τι αφορά την ε, Ρωσία, Δεδομένου των ε, ειδικών σχέσεων που έχει η Κύπρος με τη Ρωσία, χρηματοοικονομικών, ε, τουριστικών σχέσεων κλπ. Νομίζω ότι η Κύπρος θα, θα είχε κάποια ιδιαίτερη άποψη σε ό,τι αφορά των οικονομικών και εμπορικών, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δυσκολίε που απορρέουν από το γεγονός ότι η, η Ρωσία ενισχύει τις εμπορικές οικονομικές ε, σχέσεις Ταλωνιακής Ένωσης με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία και αντίστοιχα απορρέει ότι και ζητά από την Ένωση να συμμετάσχει πιο ενεργά στη λεγόμενη ευρωασιατική κοινότητα αντί να συνδέεται άμεσα με μας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί αυτή την μεταστροφή και να αρχίσει να διαπραγματεύεται άμεσα με την Ευρωασιατική Επιτροπή αντί με την Ρωσική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα αρχικό ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε απαντήσει, δεν έχουμε λάβει απάντηση ακόμα από το Συμβούλιο και είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό, όχι μόνο από άψη πολιτικής αλλά και από άψη εμπορικών σχέσεων. Δεύτερον, κάτι με το οποίο δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την Κυπριακή Προεδρία ήταν το θέμα της, ε, του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά. Δηλαδή, η, η καταληκτήρη ημερομηνία για τις χώρες ε, ΑΚΕ για να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφορετικά θα χάσουν το προτιμησιακό καθεστώς που έχουν στα πλαίσια των συμφωνιών του Κοτονού. Μετά την ψηφοφορία που έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που άλλαξε την καταληκτήρια προθεσμία από το 2014 στο 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντί να αναζητήσει κάποιο συμβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να τηρήσει την ε, άκαμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως εκ τούτου να κλείσει την πιθανότητα μιας ε, πρώιμης ε, συμβαστικής λύσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο το Συμβούλιο επέλεξε αυτή τη λύση. Αντί να προσπαθήσει να έχει μια πρώιμη ε, συμβαστική λύση μεταξύ των τριών οργάνων. Και νομίζω ότι η απόφαση αυτή προκάλεσε τελικά καθυστέρηση για τη λήψη μιας απόφυσης η οποία χρειάζεται. Γιατί βέβαια οι αφρικανικές χώρες, οι αφρικανικές εταιρείες, οι εισαγωγικές, εξαγωγικές εταιρείες και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν πολύ νωρίτερα με τι θα έχουν να κάνουν και τι καθεστώς θα αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να προτείνετε κάτι σχετικό στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία για να βρεθεί ένας λογικός συμβασμός μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων το νωρίτερο δυνατόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κίνα. Ασπαστήκατε την απόφαση της ε, Επιτροπής να υπάρξει μια συμφωνία επενδύσεων με την κοινωνία που δεν θα φορά μόνο την προστασία των επενδύσεων αλλά και τα θέματα πρόσβασης στην αγορά. Το πρόβλημα το οποίο διαβλέπω εδώ είναι το κατά πόσον το Συμβούλιο έχει αντιμετωπίσει το θέμα ότι εάν υπάρχει και μία διάσταση πρόσβαση στην αγορά, κατά η συμφωνία αυτή θα έχει και ένα κεφάλαιο περί αηφόρου ανάπτυξης και ρήτρα περί σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτή είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όλες οι συμφωνίες που αφορούν πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να μην έχουν και αυτές τις διαστάσεις. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να έχουμε μια τέτοιου είδους συμφωνία και με αυτές τις ε, δύο διαστάσεις και θα μπορούσε ή ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απεμπολίσει την αναζήτηση, την επίτευξη αυτών των δύο στόχων, των δύο διαστάσεων, προκειμένου να συνάψει τη σχετική συμφωνία με την Κίνα. Τώρα, Μερκοσούρ, περιοχή Μερκοσούρ δεν αναφέρεται κάτι σχετικά με τη συμφωνία. Δεν είναι δύσκολο βέβαια να κατανοήσουμε το γιατί δεν αναφερθήκατε, γιατί απλώς δεν συνέβη και τίποτα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Πώς ε, αποτιμάτε την κατάσταση πώς βλέπετε και πώς αποτιμάτε την έλλειψη πρόοδου στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ και ποια είναι η αψία σε ό,τι αφορά τις συνέπειες για τις χώρες που είναι τόσο αντίον, αν θέλετε, του εμπορίου, όπως η Βολιβία και το Εκουαδόρ που έχουν ενταχθεί στην Συμφωνία Μερκοσούρ το θεωρείτε δυνατό και πιθανό να υπάρξουν σοβαρές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Τέλος, θεωρώ γενικά ότι η Προεδρία σας ήταν ε, επιτυχές, που αυτό για μια τόσο μικρή χώρα είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην ποιότητα της ε, προεδρία που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη τους και χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαι ευτυχή που μια τόσο μικρή χώρα που για πρώτη φορά αναλαμβάνει την ε, Προεδρία και όντας την ε, περιφέρεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να προσφέρει, να αποδώσει τόσα πολλά. Ποια θα ήταν λοιπόν η σύστασή σας στην επόμενη Προεδρία που ακολουθεί γιατί ακολουθούν και οι πρώτε προεδρίες μικρών χωρών, των βαλτικών χωρών που θα ακολουθήσουν. Ποια θα είναι η σύστασή σα, λοιπόν στις χώρες αυτές. όταν θα αναλάβουν αυτές με τη σειρά τους Προεδρία του Συμβουλίου. Τι θα μπορούσατε να τους πείτε, ώστε να είναι εξίσου επιτυχής όσο και η Κύπρος. Ποιο είναι το κλειδί δηλαδή για μια μικρή χώρα, προκειμένου να είναι επιτυχής στην ανάληψη της ε, Προεδρίας της ε, Ένωσης. Έχω άλλο ένα αίτημα. Κριστιαν Μουσκαρτίνη. Μουσκαρτίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ως ε, Ευρωβουλευτής είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Κύπρο πριν από κάποια χρόνια και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια που κατέβαλε η Κυπριακή Προεδρία τους μήνες, αυτός, τους μήνες αυτούς. Ε, παραμένουν όμως ε, κάποια ερωτήματα που θα ήθελα να απευθύνω στην Προεδρία αυτή, ελπιστώντας ότι η Προεδρία αυτή θα μπορέσει να τα διαβιβάσει και στην επόμενη Προεδρία για να αντιμετωπίσει δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά συνεχίζει να αντιμετωπίζει και να έχει διμερείς ε, συμφωνίες και σχέσεις με τρίτες χώρες. Γνωρίζουμε όμως ότι στο μέλλον η δημοκρατία και η ειρήνη στον κόσμο θα συνδέονται και με το σεβασμό των κανόνων που θα πρέπει να διέπουν και να περιορίζουν τα διάφορα αντίστοιχα τρίτα κράτη. Και όταν ευελπιστώ σύντομα έχουμε ενδεχομένω μια συμφωνία με την Ινδία, όταν η Ινδία έχει επιδείξει ότι δεν ε, σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες μέχρι στιγμής και μέχρι στιγμής κρατά φυλακισμένους δύο ε, Ιταλούς αξιωματούχους, που το μόνο τους αδίκημα ήταν ότι διέπραξαν το καθήκον τους σε διεθνή χωρικά ύδατα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να θέσει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείξει αλληλέγγυα όχι μόνο στην Ιταλία ως Ιταλία, ως κράτος μέλος, αλλά αλληλέγγυα σε οποιονδήποτε δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ε, εκείνων που δεν σέμβανται ε, τις ε, αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά χωρικά ύδατα κλπ. Δεύτερο ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποτέ δεν εξέτασε τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τον ορισμό και την ονομασία των προϊόντων η, σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον κανονισμό αυτό τον Οκτώβριο του 2010. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως τον απέσυρε και οι Ευρωπαίοι πολίτες έμειναν κατά βάση οι, μονοι... στον κόσμο που δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των εμπορευμάτων που αγοράζουν από τρίτες χώρες. Αυτό το δικαίωμα το έχουν οι Κινέζοι, το έχουν οι Ινδοί, το έχουν οι Αμερικανοί, το έχουν οι Μεξικανοί, οι Καναδοί όχι πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι, κανόνες που διέπουν το, ευρω, το διεθνές δίκαιο ή ε, ισχύουν για τους πάντες ή για κανέναν. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ la ε, η προσέγγιση και ο σεβασμός. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλειφθεί ως μια χώρα, αν θέλετε, ως, ως μια πολύ σημαντική ενιαία εσωτερική αγορά, θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες αυτές. Και το Συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει σχετικά το αίτημα του Κοινοβουλίου. Δεν λέω ότι το Συμβούλιο πρέπει απαραίτητα να συμπανταχθεί με την γνώμη του Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να ανοίξει τουλάχιστον ένα άτυπο διάλογο και να το αντιμετωπίσει το θέμα. Αντίθετα δεν υπήρξε αυτό ο διάλογο και δεν υπήρξε καμία αντιπαράθεση και Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απέσυρε την σχετική τροπολογία. Θέλουμε κάποια σχετική ε, απάντηση στα θέματα αυτά, τα οποία μας είναι τόσο σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε μια πληθώρα ερωτημάτων να απαντήσετε. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την απάντηση που θα δώσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να ξεκινήσω με τα ερωτήματα ε, της κυρίας Κέλλερ. Να πω ότι ε, είπα και στην ομιλία μου ότι στην, η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά βρίσκεται στα τελικά σταδιά. Είναι αλήθεια ότι ενώ επιτεύχθηκε σημαντική προοδός υπάρχουν προβλήματα σε σχέση ε, κυρίως με τις εξαγωγές γεωργικών και χτινοτροφικών προϊόντων όπως αναφέρεται. Να πω ότι πρόσφατα έγινε συνάντηση του Επίτροπου Ντεγούχτ με τον Καναδό ομόλογο. Μάλιστα στη συνάντηση ήταν παρόν και ο Επίτροπος ε, Γεωργίας ε, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα και εύχομαι και ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα διοντηρώντας βεβαίως κυρία Κέλλε και πρέπει να σας διαβεβαιώσω αυτόν αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε από την Επιτροπή τις βασικές αρχές ε, σε ό,τι αφορά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρώ και με τη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο ότι θα ξεπεραστούν όπως αναφέρεται οι κόκκινες γραμμές, ε, κάποια ζητήματα που βεβαίω είναι απέτηση του Καναδά. Το δεύτερο θέμα που αφορά τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είπα και στη συνάντησή μας εδώ τον περασμένο Ιούλιο ότι ως Προεδρία, σεβόμενη την απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, δεν προχωρήσαμε στο θέμα, αναμένοντας βεβαίω και την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα έλεγα ότι υπάρχει μια παγωποίηση στο θέμα. Ε, και ελπίζω ότι ε, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρουν τον τρόπο ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι διαφωνίες που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία, α, δεν θεωρώ ότι άλλαξε ενουσιοδός η διαπραγματευτική εντολή. Δίθετα, έχουμε μπει όλοι και στη συζήτηση που είχα εδώ τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες οσορροπίες, όπως ανάφερα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε σε κάποιους ευαίσθητους τομείς τα ενδιαφέροντα και τα εμπορικά συμφέροντα κρατών μελών και είναι εδώ που βρήκαμε ακριβώς ε, τη συμβαστική λύση. Από τη μια δίδοντας τις διαπραγματευτικές εντολές να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, που είναι τόσο σημαντικές για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την άλλη ε, να θέσουμε εκείνα τα ζητήματα που είναι ευαίσθητα για κάποια ε, κρατημέλη ώστε να μπορέσουμε να ξεπερνούσαμε τα διέξοδο και αυτή είναι τη λύση που βρήκαμε στο τελευταίο ε, ε, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Σύνθεση Υπουργών Εμπορίου στις 29 Νοεμβρίου. Με την ιδέα εκείνο που θα έλεγα είναι ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα. Επιθυμία του Συμβουλίου είναι να καταστούν οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες για εξέβρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ανατονίσει. ε, η προσπάθεια μας υπάρχουν προβλήματα σε πάρα αρκετούς ε, τομείς όμως εκείνο που έχω πει ότι ε, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση πριν από μερικούς μήνες ε, και η προσπάθεια μας είναι να ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες βέβαια στο το 2013, αλλά εκείνο που έκφρασα με την τοποθέτησή μου είναι την βούληση της, ε, ε, του Συμβουλίου να προχωρήσει και εδώ επειδή αναφέρομαι στην Ιδία ε, θα ήθελα να τονίσω ξανά επειδή αναφέρθηκε η κυρία Μεσκαντίνη για το θέματα του, το πόσο μια χώρα σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες, ε, κυρία Μεσκαντίνη είναι απαραίτητος όρος ότι εκεί που συνάπτουμε συμφωνίες πρέπει να σέβονται τους διεθνούς κανόνες και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπα και στην εισαγωγή μου παρέμβαση, το είχα, το, είχα τοποθετηθεί και στην άξη της Προεδρίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο. Δεν είναι μόνο θέματα αλληλεγγύης μεταξύ ε, των κρατών μελών και αλληλεγγύης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κράτη-μέλη και πολίτες της είναι υποχρέωση απέναντι σε κανόνες ε, του διεθνούς δικαίου απέναντι στο σεβασμό ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και το σεβασμό απέναντι στις, ε, ε στις αρχές των, των διεθνών συμφωνιών. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ε, Σιγκαπούρης, να πω ότι εκείνον καταλήξαμε σε αυτές τις ε, συμφωνίες. Ε, αναμένεται αυτό να αποτελεί σημείο μία και άλλα. Ε, καταφέραμε ένα νέο αλλά σημαντικό στοιχείο στι διαπραγματεύσει με τη Σιγκαπούρη ήταν η επιδίωξή μας για συμπλήρωση συμφωνία ενό περιεκτικού πράσινου πακέτου, προκειμένου να μπορεί να προωθούν ε, νέες ευκαιρίες σε τομείς ε, πράσινας ανάπτυξης ε, και έχετε δίκιο κύριε Κέλλερ ότι είναι εδώ μέσα από τους μηχανισμούς που θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε ώστε να είναι πιο αποφασιστική συμμετοχή, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ε, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα του Προέδρου του κυρίου Μορέιρα. Πρώτα-πρώτα, αγαπητέ καθηγητέ, να πω ότι ανεξάρτητα από, από τις ειδικέ σχέσεις που έχει η Κύπρος ε, και σε αυτόν τον τομέα όπως σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας λειτουργήσαμε ως Προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακριά από οποιασδήποτε εθνικές επιδιώξεις ή εθνικά ζητήματα που είχαμε ε, μπροστά μας. Ε, γι' αυτό δεν τοποθετηθήκαμε ή τοποθετούμαστε ε, γύρω από αυτό το θέμα στη βάση αυτών των σχέσεων. Εξάλλου και στην εισαγωγή μου παρέμβαση είπα ότι είναι σημαντικό και αυτό συζητήσαμε και στο τελευταίο Συμβούλιο να είναι συνεπής η Ρωσία α, στις διεθνείς συμφωνίες, στις πολυμερείς ε, σχέσεις για να μπορέσουν να προχωρήσει ε, οι σχέσεις μας ε, με τη Ρωσία να μην παραβιάζονται δηλαδή και οι όποιες σχέσεις. Ε, πρέπει να πω ότι ε, θεωρούμε ότι σημαντικό ότι η Ρωσία εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τώρα, σε σχέση με την Ελληνική ε, Ένωση ή τι ελληνικέ σχέσει τη Ρωσία με Λευκορωσία και το Καζαστά, ναι, είναι, θεωρώ και εγώ, κύριε Μωρέρα, ότι είναι ένα θέμα αυτό, το σε ποια βάση θα μπουν οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν μπορούμε προ το παρόν να δεχτούμε ε, ε, τη διαπραγμάτευση με την Ευρωασιατική Ένωση ε, εφόσον οι χώρες, οι, χώρες της δεν είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου άρα επιδίωξή μας είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τη Ρωσία. Για τον κανονισμό που αφορά την πρόσβαση στην αγορά το Συμβούλιο έχει προχωρήσει στη ε, ε, σύναψη σύμφωνα σε ό,τι αφορά το κείμενο της προσκαμισμού, οδηγώντας ουσιαστικά τις διαδικασίες στη δεύτερη άγνωση. Οι ε, ενέργειες του Συμβουλίου βεβαίως αντανακλούν την υποστήριξή μας προς την πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ουσιαστικά έχει υιοθετήσει την πρόταση με μια τεχνική προσαρμογή ώστε να ληφθεί υπόψη η επικύρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομική εταιρικής σχέση τη, από τη Ζιμπάμπουε Πιστεύει το Συμβούλιο ότι ε, η θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποτελεί έναν ισορροπημένο ε, ε, σύνολο και είναι εδώ που προβλέπεται να υπάρξουν επικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάδοση και πρέπει να πω καθηγητέ ρε ότι υπήρχε ομοφωνία στο Συμβούλιο. για τα θέματα της αυτό που θα ε, συμβουλεύαμε ε, την Ελλαδική Προεδρία είναι να προχωρήσει σε αυτήν τον διάλογο ε, με πνεύμα συμβασμού ώστε να εξευρεθεί η λύση και να προχωρήσει στο θέμα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα για την Κίνα και την για τη Συμφωνία Επενδύσεων, την οποία συζητήσαμε, θα έλεγα, αρκετά διεξοδικά στο τελευταίο Συμβούλιο στις 29 ε, Νοεμβρίου. Ε, νομίζω δεν υπάρχει καμία αφορία ότι η Κίνα είναι ένα σημαντικός στρατηγικός εταίρος ε, και οι όποιε ενέργειες για συνεργασία και βάθηση των εμπορικών μας σχέσεων είναι θεμητές και επιθυμητές. Αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα προσφέρει περισσότερα ωφέλη από τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει αρκετά κρατημέλη με την Κίνα. Ε, από την συζήτηση που έχουν γίνει για την Προεδρία μα, τόσο σε υπουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, θεωρώ ότι υπάρχουν οι προποθέσει για έναρξη των διαπραγματεύσεων στο προσεχέ μέλλον. Ε, Ακόμα δεν έχει γίνει πρόταση από την Επιτροπή ενώ στι λεπτομέρειε τη για, για, να περιληφθούν, για να ληφθούν υπόψη ε, τα δύο ζητήματα που έχετε θέσει σε σχέση με την ε, εφόρον ανάπτυξη ε, και την ανθρώπινα δικαιώματα. το Συμβούλιο υιοθέτησε, όπως γνωρίζετε, τον περασμένο Ιούνιο των στρατηγικών πλαίσιων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς όρους και θεωρώ είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τα θέματα της Σουρ έχετε δίκιο καθηγητή Ρέιρα, το ότι δεν αναφέρθηκα αποτυπώνει και μια κατάσταση η οποία είναι στάσιμη. Ε, δηλαδή δεν υπάρχει πρόοδος. Και αυτόν επηρεάζουν αρνητικά ε, το είπαμε και στη συζήτηση όταν, τον Ιούλιο όταν ήμουν εδώ ε, στην Επιτροπή σας ε, οι εξελίξεις στην Αργεντινή. Όμως πρέπει να πούμε ότι η Σου δεν αποτελείται μόνο από την Αργεντινή αλλά και από άλλους στρατηγικούς εταίρους. Για παράδειγμα η Βραζιλία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προδυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση των προβλημάτων προκειμένου να δοθεί μελλοντικά νέα προοπτική στην ευβάθυνση και εξομάλυνση των προηγούμενων μα σχέσεων με τις χώρες του Μερκοζού. Ε, τα μέτρα προστατευτισμού που έχει πάρει η Αργεντινή προκαλούν σημαντικές ανησυχίε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς παρακολουθούσαμε στενά τις εξελίξεις, υποστηρίζουμε τις ενέργειες ε, της Επιτροπής τόσο σε διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο για αντιμετώπιση του προβλήμα, αλλά επαναλάβω πρέπει να βρούμε τους τρόμους για να προχωρήσει η συζήτηση με την Μερκεζού. Ε, στα θέματα που έθεσε η, ε, η, η κυρία Μεσκαντίνη, ε, πέρα δηλαδή από τα θέματα της Ινδίας, ε, αναφέρθηκε στο ε, κανονισμό σήμανση προϊόντων. Ε, έχετε δίκιο κυρία Μεσκαντίνη, αλλά πρέπει να πω ότι η αλήθεια είναι ότι οι αντιθέσεις στο Συμβούλιο είναι τόσο μεγάλες που όσο και αν προσπαθούμε ή προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε ως ένας μεσολαβητής, ένας, για να εξευρεθεί συμβασμός, Τελικά ε, δεν υπήρξε αυτός ο συμβασμός. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν δεύτερες ε, σκέψεις από κράτη-μέλη διότι έχετε δίκιο. Είναι ένα μεγάλο ε, κενό και πρέπει να αναγνωρίσουμε, είναι ένα μεγάλο κενό, δεν υπάρχει αυτή η σήμαση. Βεβαίω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα από του λόγου απόσυρση τη πρόσφατη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν και η πρόσφατη γνωμάτευση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που καθιστούσε την πιθανή εφαρμογή τη λόγω πρόταση μη συμβατέ με του κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. πάση όμω περιπτώσει, η συμβολή και στην επόμενη Προεδρία και στην Επιτροπή είναι να καταβληθούν όλε οι προσπάθειε ώστε να ξεπεραστούν ε, τα προβλήματα. Ε, ήθελα να ε, ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μωρέιρα πρώτα-πρώτα για τα καλά του λόγια σε ό,τι αφορά την Προεδρία και την Κυπριακή Προεδρία και ακριβώς αυτό που ήθελα να αναφέρω αγαπητέ κύριε Πρόεδρε ε, πως ε, μικρές χώρες ε, στην περιφέρεια καταφέρνουν να προωθήσουν. Και όντω ε, ε, διεκπαιρώθηκε ένα μεγάλο όγκο δουλειά και δεν αναφέρομαι μόνο στου 36 φακέλου, αναφέρομαι ότι υπήρξαν δύσκολα θέματα. Εκείνο που ήταν το πιο σημαντικό είναι ότι η Κυπριακή Προεδρία λειτουργήσε, όπως είπαμε και από την αρχή, ως ένας έντιμος και αξιόπιστος διαμεσολαβητής. Και θέλω να ευχαριστήσω βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη που αναγνώρισαν αυτόν τον ρόλο και πολλέ φορέ οι συμβαστικέ μα προτάσει γινόταν αποδεχτές ξεκινώντα με το δεδομένο ότι μια μικρή χώρα δεν έχει να εκπροσωπήσει ε, μεγάλα συμφέροντα ή πολλέ φορέ ε, άλλα ε, εθνικά συμφέροντα που πολλέ φορέ μπορεί να επηρεάζουν το να ασκήσει κάποιο την Προεδρία ω ένα πραγματικά κρίκο, ένα έντιμο διαμεσολαβητή. Το δεύτερο ότι υπήρχε σημαντική επαφή και συνεχής επαφή με όλα τα θεσμικά όργανα. Να σας θυμίσω, ε, καθηγητή Μωρέρα, ότι στην πρώτη μας συνάντηση ε, πριν να λάβουμε την Προεδρία όταν επισκεφθήκατε την Κύπρο είχαμε πει τότε στην ομιλία ότι θα πρέπει πολλές φορές ξεπερνώντας ε, τι α, τις που υπάρχουν και τους κανόνες ότι πρέπει πρώτα πρώτα να συζητούμε και όταν υπάρχει μια συμφωνία να έρχεται ω τελικό προϊόν για να τοποθετεί το Ευρωκοινοβούλιο και ότι θα μπορούσε και αυτό είναι θέμα πολιτική βούληση να βρεθεί η φόρμουλα να υπάρχουν συνεχεί επαφέ. Δηλαδή, πριν να καταλήξει η Επιτροπή και το Συμβούλιο σε μια θέση, να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θέσει του Ευρωκοινοβουλίου. Που θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά, είναι από τα θεσμικά όργανα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες, στους προβληματισμούς και στους ανάγκες τους. Και τέλος, θεωρώ σημαντικό ότι όταν υπάρχει ε, λίγη, είναι λίγη η λειτουργή μας, αλλά ε, οι λειτουργοί μας λειτουργήσαν πολύ ε, εντατικά και είναι κλειδί για μια προεδρία, ο προεδρεύω, να έχει άμεση και καθημερινή επαφή με όλους τους ανθρώπους που διεκπαιρώνουν τους φακέλους και την πολιτική. Και εδώ πιστεύω είναι το κλειδί της επιτυχίας ε, το ε, μικρό ε, χωρών και θέλω να πω ότι για μας ως Κύπρος μας έδωσε μια, ήταν μια τεράστια εμπειρία, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω και εσάς και το Συμβούλιο και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να διεκπαιρέσουμε αυτούς τους φαγγέλους. Εξάλλου, στο επίκεντρο της προσοχής μας και στην έννοια όλων μας είναι να δουλέψουμε ιδιαίτερα στι σημερινέ δύσκολε συνθήκε για την Ευρώπη, για μια καλύτερη Ευρώπη όπω ήταν και ο στόχο τη Κυπριακή Προεδρία, μια καλύτερη Ευρώπη ιδιαίτερα ε, για του πολίτε τη. Σα ευχαριστώ και πάλι. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το ενδιαφέρον σας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να βασιστούμε σε εσάς και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή Εμπορίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε εσάς προσωπικά και στη χώρα σας. Κυρίες και κύριοι, ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία, στις ψηφοφορίες μάλλον.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 για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα. 11 και 12 μαζί. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Υπάρχει μόνο ένας κατάλογος ψηφοφορίας που αρχίζει με τη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. πέραση της φοφορίας. Δεκτή. Η τροπολογία 5. Τροπολογία 3. Όχι. Α, είχα είχα έναν άλλο κατάλογο στα χέρια μου, λέει ο πρόεδρος. 6. Ψηφίζουμε την 6. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ε, yes, one minute or two minutes. Ένα ή δύο λεπτά λέει ο πρόεδρος απαντώντας ένα σχόλιο εκτός μικροφώνου που δεν ακούστηκε. Well, since, since is a Δεδομένου ότι είναι ένας φάκελος και ο εισηγητής θα μπορούσατε να ακολουθήσετε την, τον κατάλογο ψηφοφορία σύμφωνα με τον εισηγητή, πιστεύω. Λέει ο πρόεδρος. Μπορεί κάποιος να δώσει στους σοσιαλιστές και δημοκράτες τον κατάλογο, παρακαλώ, της ψηφοφορία ψηφοφορίας στον εισηγητή. Α, εντάξει, εδόθη και συνεχίζουμε. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ Κα... ηλεκτρονικός έλεγχος 10 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας Α, απερίφθη, απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2. Σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα τη συμβιβαστικής 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16. Ψηφίζουμε 16 πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Το δεύτερο έχει αποσυρθεί, άρα υπάρχει μόνο ένα τμήμα. Το πρώτο λοιπόν, τέλος πάντων, ψηφίζουμε τη 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μόνο μέλη μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικό έλεγχο, όχι βοηθή. 24. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 25 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή, δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 36 όχι, καταπίπτει. Σαράντα, υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. Σαράντα ένα. Υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 42. Υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. τρία, Υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. 45 υπέρ 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. γιατί, να, γιατί να ελέγξουμε, τέλο πάντων, ελέγχουμε την 56, ηλεκτρονικά 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 προς 1. Προ, προτείνω, προτείνω πρόστιμο, λέει ο πρόεδρος, για άχρηστη πρόταση ηλεκτρονικού ελέγχου. Λοιπόν, προχωρούμε. 57 ε, υπέρ κατά που έχει 58 υπέρ κατά υπέρ υπέρ 58 κατά αποχές δεκτή 58 έλεγχος ηλεκτρονικός παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας 24 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και τον δύο γνωμοδοτήσεων, ο οποίος δεν είναι σήμερα μαζί μας, ε, λείπει στο εξωτερικό σε μια πολιτική αποστολή, πολιτικής φύσης. Προχωρούμε στο 13 του Ντάνιελ Κασπάρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στο σημείο 10... Ένα λεπτό λέει ο να βάλω τα ακουστικά μου. Πριν προχωρήσουμε στο, ψηφοφορία για το 13, θέλω να διευκρινίσω ένα στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει όλους. Μία χώρα την οποία αφορά αυτή η ψηφοφορία είναι η Ζιμπάμπουε και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολη στη Ζιμπάμπουε και γι' αυτό προτείνω ταυτόχρονα με αυτή την έκθεση να παρουσιάσουμε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο όπου ε, θα εστιάζουμε ξανά ως Κοινοβούλιο στη στην κατάσταση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις ανησυχίες που έχουμε για το λαό της χώρας αυτής. Και ε, πιστεύω ότι θα με υποστήριξετε όλου σε αυτό το ψήφισμα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Φρανσέσκα Κέλλερ. Και εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα. Θα ήθελα να τη διευρύνω λιγάκι, διότι η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ανέφερε και άλλα επιχειρήματα ότι το θέμα αυτό δεν συνδέεται μόνο με τη Ζιμπάμπου, αλλά μπορούμε να το διευρύνουμε λιγάκι και για άλλες χώρες. Δεν σας αρέσει? Όχι. Εντάξει, εμείς αυτό θα προτείναμε. Ευχαριστώ πάντως. Ο κύριος ε, Ρόμπερτ Σέρντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους Βρετανούς, μακροχρόνιο πρόβλημα και βεβαίως ολόθερμα υποστηρίζω αυτό που είπε ο Ντάνιελ. Είναι ένα μεγάλο, πολύ ανησυχητικό πρόβλημα και εμείς έχουμε αποφασίσει να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα διότι μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι κατάσταση στη Ζιμπάβουε και θα βοηθήσουμε και στη σύνταξη του ψηφίσματος. Ο κύριος Κούτας. Και εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση του Ντάνιελ και περιμένουμε τον Ιανουάριο να συζητήσουμε το θέμα. Πολύ ωραία. Έτοιμοι για την ψηφοφορία λοιπόν και συμφωνούμε για το, την υποστήριξη του ψηφίσματος όπως εισηγήθηκε ο εισηγητής, Ντάνιελ Κάσπαρη. Ας ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Ένα και δύο, ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται και ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος όπως δεν τροποποιήθηκε. Ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Α, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Και εγκρίθηκε με 20 υπέρ 5 κατά μία αποχή. Ωραία, προχωρούμε στο 14. Προφορική ερώτηση για ε, το, την ε, προέλευση ε, ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. 14. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή προφορική ερώτηση. Θα ψηφίσουμε την ίδια ερώτηση ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Οι ερωτήσεις μας προς το Συμβούλιο δεν γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνουν δεκτές ως αίτημα για τη δήλωση του Συμβουλίου. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι διαδικαστικά οι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο δεν γίνονται δεκτές, γι' αυτό θα αλλάξουν φύση και θα είναι προφορικές ερωτήσεις για τη δήλωση του Συμβουλίου. Τώρα ψηφίζουμε προφορική ερώτηση της Επιτροπής προς την Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι το 14, είναι το 14. Ήδη προφορική ερώτηση, αλλά προς την Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεκτή, λοιπόν, η ερώτηση ομόφωνα με 26 ψήφους. Α, ξέχασα να σας πω το προηγούμενο αποτέλεσμα της προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο, δηλαδή προς τη δήλωση ήταν 24 υπέρ, 5 κατά μία εποχή. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα στο 15. Είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα, για την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο της προσχώρησης τους. Ο κύριος Βίνκλερ μου επιτρέπετε πρόεδρε ένα διαδικαστικό, διαδικαστικό ερώτημα που γενικό όχι μόνο σε αυτό το σημείο. Κάτω-κάτω στην, ε, στον κατάλογο ψηφοφορίων λέει ότι το υιοθετημένο κείμενο μπορεί να υποστεί αλλαγές για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή δεν βλέπω ποιο είναι το νόημα αυτής της υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας. Τι θα πει τεχνικές προσαρμογές, εμείς δεν έχουμε ε, τροπολογίες, δεν έχουμε τίποτα. Τι σημαίνει αυτή η υποσημείωση. Ο πρόεδρος, να σας καθησυχάσω, είναι καθαρά τεχνική διαδικασία που γίνεται πάντοτε. Είναι μία σημείωση και η διατύπωση αυτή ανταποκρίνεται στα τεχνικά πρότυπα. Δεν δίνεται καμία εξουσιοδότηση για ουδεμία αλλαγή. Είναι απλώς ένα γλωσσικό νομικό θέμα και σε κάθε φάκελο υπάρχει αυτή η υποσημείωση. Ακόμα και σε κανονισμούς που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, Κοιτάξτε κύριε Βίνκλερ, θα ελεγχθούν, θα ελεγχθούν από εμάς πριν υιοθετηθούν επισήμως. Πάντοτε θα υπάρχει ένας έλεγχος εάν ε, συνάδουν με τις ε, γλωσσικές νομικές διαδικασίες. Εδώ δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, καμία ε, επιπρόσθετη εξαίρεση εδώ δεν προστίθεται με αυτή την υποσημείωση, απλώς είναι μια ε, στάνταρ πρότυπη διαδικασία αυτή, τεχνικής φύσεως. 15 λοιπόν. Προχωρούμε στο 15. Σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Πέρασε ψηφοφορίας. Η Εγκρίσκε με 25 ψήφους υπέρ μια αποχή. Και τώρα... An item which was added to our agenda. Προσθέθηκε στην η ημερήσια διάταξη μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την παρούσα κατάσταση των ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων με το Μερκοσούρ. Ε, ψηφίζουμε την προφορική ερώτηση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, δεκτή ομόφωνα 24 ψήφοι. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Και ας προχωρήσουμε στο θέμα, στο 16. Θα ήθελα να σας ζητήσω να παραμείνετε μαζί μας και θα μας λείψετε πολύ. Έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που αξίζει να τον ε, παρακολουθήσουμε. Το επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο Doing Business 2013. Επιχειρήν δηλαδή 2013. Μπορώ να έχω την προσοχή σας. Παρακαλώ πολύ όσοι αποχωρείτε, πράξτε το με ησυχία και όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Μην αρχίζετε διαλόγου και συζητήσει με στην αίθουσα. Και αυτό βέβαια ισχύει όχι μόνο για το προσωπικό, αλλά και για τα μέλη της Επιτροπής. Το επόμενο θέμα λοιπόν, όπως σας είπα, πραγματεύεται την ε, έκθεση επιχειρήν 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση σας παρουσιάζω τον ειδικό προσκεκλημένο, τον κύριο Αγκούστο Λόπεξ Κλάρος, ο οποίος είναι διευθυντής ε, της ε, ομάδας ανάλυσης παγκόσμιων δικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας από το Μάρτιο του 2011. Ο προσκεκλημένος μας ε, προηγουμένως ε, ήταν επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής του προγράμματος Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Και πριν το φόρουμ, πριν έρθει στο φόρουμ, δούλεψε για τους Lehman Brothers και το Διεθνές Ταμείο και ήταν καθηγητής ε, οικονομικών στο Πανεπιστημίο της Χίλης του Σαντιάγκο. Είναι ο συντάκτης πολυάριθμων ε, άρθρων και δημοσιεύσεων σε ό,τι αφορά διεθνή χρηματοοικονομικά ζητήματα. Θα μας παρουσιάσει την πρόσφατα δημοσιευστής ετήσια έκθεση του Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Επιχειρήν 2013. Έξυπνοι κανονισμοί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Uh, and have a with him. Θα ακολουθήσει και συζήτηση μαζί του. Ε, αυτή η ετήσια έκθεση ε, βαθμολογεί τις παγκόσμιες οικονομίες σε διάφορους δείκτες, ε, όπως ε, την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητα, την επίλυση του πτωχευτικό δίκαιο και την επίλυση αξιόχρεων και το επιχειρήν διασυνοριακά. Με πολύ μεγάλη ευχαριστήσεις θα σας ακούσουμε σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση καονιστικών εμποδίων σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα και επιχειρηματικό κλίμα και την σχετική βαθμονόμηση χωρών όπως είπα η Κίνα, η Ρωσία κλπ. σε ό,τι αφορά την ε, παγκόσμια επιχειρηματικότητα. Σας καλωσορίζουμε στην ε, παρουσίασή μου στη συνέλευση της ε, Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο, ένα 15 και μετά θα ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να παρουσιάσω τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης επιχειρήν 2013, ένα κοινό project της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας και του ε, Διεθνούς ε, Χρηματοοικονομικού Οργανισμού. Όπως ξέρετε, την τελευταία δεκαετία στον Παγκόσμια Τράπεζα και στο IFC έχουμε αναπτύξει μια σειρά δικτών που ε, αποτυπώνουν διάφορες διαστάσεις του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Για πάρα πολλά χρόνια η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιούσε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο με τίτλο «Έρευνες επιχειρήσεων» που χρησιμοποιούμε σε... και παρακολουθούμε κάπου 130 χώρες όλο τον κόσμο. Στις επισκοπήσεις αυτές τις έρευνες προσπαθούμε να μετρήσουμε την επιχειρηματική κοινότητα σε ό,τι αφορά ποιε είναι τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά το επιχειρήν και το επενδυτικό κλίμα στις ε, καθημερινές τους δραστηριότητες, στη δημιουργία δηλαδή νέων θέσεων απασχόλησης και συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτές οι επιχειρηματικές ε, έρευνες, έρευνες της επιχειρηματικότητας, μας έχουν δώσει πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σε ό,τι αφορά κάποια διέξοδα που υπάρχουν, κάποια στενέματα αν θέλετε, και στη διεθνή οικονομία, αλλά και στις βιομηχανοποιημένες χώρες και στον απτυσσόμενο κόσμο και στις βιομηχανικές χώρες. Ξέρουμε για παράδειγμα το θέμα της φορολογίας είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολύ σημασία αν είναι τόσο πολύ οι συντελεστέ φορολόγηση που τελικά είναι αντικίνητρο για την επιχειρηματική κοινότητα ή δυνάμει επενδυτέ, στην ε, προσπάθειά τους ε, της ε, διευθέτησης ζητημάτων με τους εφοριακούς. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της φορολογίας. Το κατά πάσο αν μπορεί κάποιος να εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις εύκολα και γρήγορα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην αρτήση του χρόνου το project αυτό, το επιχειρήν δηλαδή, έχει αναπτύξει 10 δείκτες που συλλαμβάνουν διαφορετικές ε, ενδείξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προσπαθούμε για παράδειγμα να αποτιμήσουμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας για να εγγράψει στο εμπορικό επιμελητήριο την έναρξη μιας, τη δημιουργία μιας νέας Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το κόστος και τα ε, κανονιστικά ομπέδια που υπάρχουν για τις διασυνοριακέ επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Ε, προσπαθούμε να αποτυπήσουμε το κόστος και τη διαδικασία ε, καταγραφής μιας επιχείρησης και τα θέματα πνευματική ιδιοκτησίας. Κοιτούμε τα θέματα επίλυσης διενέξεων, θέματα σεβασμού εμπορικών συμφωνιών κλπ. Στην αρτήση του χρόνου έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο σώμα δικτών που δίνουμε στην έκθεσή μας αυτή, σε αιτήσια έκθεση, στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Φέτος, που είναι η δέκατη σχετική επέτειος αυτού του project, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να δούμε πιο ε, μακρόπνα τα πράγματα, να δούμε ποιες είναι οι τάσεις, ποια μαθήματα πήραμε από αυτό το ενδιαφέρον αυτό εγχείρημα και στα επόμενα λεπτά θα ήθελα να σας δώσω κάποια γενική ε, επισκόπηση των πιο, σημαντικών αποτελεσμάτων που έχουμε από το project αυτό. Κάθε χρόνο κοιτάμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκάμινου σε όλο τον κόσμο. Καλύπτουμε 185 χώρες ε, ε, και ουσιαστικά καλύπτουμε πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ με την έρευνα αυτή. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εδώ στην ε, ε, φούσκα που φαίνεται να υπάρχει στην υποσαχάρια Αφρική. Αν πάτε το 2005 υπήρχε ένα σύνολο 33% χωρών της υποσαχάριας Αφρικής που είχαν εφαρμόσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων και που ε, καλύπτονται από τους δείκτες μας. Αν δείτε τα τελευταία χρόνια, ο μέσο όρο αυτός έχει πέσει λιγότερο από 17%. Ουσιαστικά υπήρξε διπλασιασμό των χωρών υποσαχάρη ε, Αφρική που ξεκίνησαν με τα ρύθμε τις οποίε συχνηλατούμε μέσω των επιχειρηματικών δικτών και αυτό το θεωρήσαμε πάρα πολύ ενθαρρυντικό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η υποσαχάρη Αφρική έχει το πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, το πιο ε, πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο το λιγότερους συνεκτικούς ε, και συμπαγείς κανόνες που δυσκολεύει πάρα πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα σα δείξω κάποιες διαφάνειες που ε, παρακολουθούν και χλατούν κάποιους από τους διεκτήτες που έχουμε. Έχουμε έναν δίκτυ που επωνομάζεται το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Μετρά τον χρόνο, τον αριθμό διαδικασιών και το κόστος των ε, συμπαρομαρτών για την ξεκίνηση μια επιχείρηση. Το 2005 βλέπει λοιπόν κανείς ότι τότε υπήρχαν περίπου 40 ε, χώρε όπου χρειαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Αν έρθουμε τώρα στο παρόν, το 2012, έχει ανέβει ο αριθμό αυτό σε 105, δηλαδή έχουμε 105 χώρε που χρειάζεται λιγότερες από 40 μέρε να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Και η αύξηση από το 40 προς το 105 κατά κύριο λόγο σημειώθηκε στο αναπτυσσόμενο χώρο, στην υποσαχάρη Αφρική, δηλαδή στη Λατινική Αμερική, στη Νότιο Ασία. Αυτό το βρίσκουμε εξαιρετικά ενθαρρυντικό όχι γιατί ο δίκ, η δίκτυση είναι αυτός σκοπός, αλλά γιατί συνδεδεμένος με το δίκτυο αυτό ε, υπάρχει η πραγματική οικονομία, δηλαδή μια μετρήσιμη εξέλιξη στην πραγματική οικονομία. Έχουμε εμπειρική βιβλιογραφία που δείχνει ότι σε χώρε που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση, που είναι δύσκολο για του επιχειρηματίε να προσεγγίσουν την επίσημη αγορά, είναι χώρε με υψηλό επίπεδο διαφορά, με μεγάλο ποσοστό ατύπων διαδικασιών και όσο πιο εύκολο γίνεται σε μια επιχείρηση να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, βλέπουμε μείωση στο επίπεδο των άτυπων διαδικασιών και μείωση στο επίπεδο της διαφθοράς. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Και επίσης είναι πάρα πολύ λογικό. Το περιμένει κανείς από κάποια χώρα όπου οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πάρα πολύ δαπανηρές και επαχθείς, είτε θα, φοβίζονται, θα φοβούνται οι επιχειρηματίες και θα αποθαρρύνονται, και να μπουν στην αγορά ή θα αποτελέσουν κομμάτι της άτυπης οικονομίας ή θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες συμφωνίες με φοριακούς ή άλλους αξιωματούχους που επομένως θα υποθάλπτει την διαφθορά στη χώρα. Αυτό είναι το κόστος που συνδέεται με την έναξη μιας επιχείρησης και όπως θέλετε υπήρξε μείωση σε όλο τις περιοχές του κόσμου σχεδόν χωρίς εξαίρεση την τελευταία 7 αιτία. Επειδή ακριβώ δημιουργήσουμε μια πολύ ε, εντυπωσιακή τράπεζα δεδομένων τελευταία δεκαετία, μπορέσαμε να εξετάσουμε διάφορα επεισόδια μεταρρυθμίσεων στι διάφορες χώρες που παρακολουθούμε και καλύπτουμε. Σε αυτό το συγκεκριμένο γράφημα που μπορώ εντάχει να σα εξηγήσω, εξετάσαμε ε, μεταρρυθμίσεις σε χώρε που στοχεύουν στην διευκόλυνση τη ε, εισόδου στην επίσημη οικονομία. Η, η κατακόρυφη γραμμή στο μέσον είναι η μη χρονιά, όταν άρχισαν δηλαδή κάποιε μεταρρυθμίσει. Εκεί δεν βλέπουμε τη Χιλία, τη Σουηδία, το Μαρόκο, την Κένια. Και στη συνέχεια βλέπετε την αύξηση των αριθμών των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων που, που, που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Είδα ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στα πρώτα δύο χρόνια μετά, μετά την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων αυτών, σχεδόν σε όλες τις χώρες που εξετάσαμε. Και βέβαια αυτό συνδέεται και με μια σειρά των αριθμών των καταγεγραμμένων εταιριών, αλλά και ε, παρεπόμενη αύξηση των θέσεων εργασίας, που αυτό είναι το πολύ σημαντικό ε, αντιστάθμισμα και το όφελος από τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ένας άλλος δείκτης που θα σας αρέσει ιδιαίτερα, με δεδομένο την ε, φύση αυτής της Επιτροπής, ε, εξετάζουμε λοιπόν το χρόνο που χρειάζεται για να ε, υπάρξει εξαγωγή από ένα, ε, ενός κοντέινερ από τον κύριο λιμένα μιας χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και πάλι υπάρχουν εμπειρικές ε, μαρτυρίες από τη βιβλιογραφία που ε, αναφέρουν ότι για κάθε μέρα που καθυστέρησης εμπορίου ε, λόγω βιογραφειοκρατικών εμποδίων ε, και άλλων γενικών διαδικασιών, τελωνιακών διαδικασιών, για κάθε μέρα καθυστέρησης, δηλαδή αναχώρησης του κοντέινερ από ένα λιμένα, υπάρχει μείωση κατά 1% του συνολικού όγκου των ε, εμπορικής δραστηριότητα. Και αν μιλήσουμε ιδιαίτερα για τις χώρες Αφρική, Αφρικής, ε, η ελαστικότητα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη, φτάνει το 3 με 4%. Επειδή το εμπόριο ήταν ακριβώς μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης στη μεταπολεμική περίοδο, είναι σημαντικό να δούμε ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να εξαχθεί ένα κοντέινερ έχει μειωθεί σε όλα τα σημεία του πλανήτη, σε κάθε περιοχή που καλύπτει η μελέτη τη Παγκόσμια Τράπεζα. Και το δεύτερο κομμάτι που βλέπετε στο, η στήλη, στο γράφημα αυτό, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και πάλι βλέπουμε σημαντική ε, μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξαγωγή ενός κοντέινερ. Εδώ έχουμε καταβάσει την ίδια ιδέα, αλλά με έναν άλλο δείκτη, που είναι ο δείκτης ε, των καταβεβλημένων φόρων. Δηλαδή, ε, καταγράφουμε και τον όγκο των φόρων που ε, εισπράττονται, αλλά και τον χρόνο που χρειάζεται για τη φορολογική διεκπαιρέωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλο τον πλανήτη, σε κάθε περιοχή συμπεριλαμβανομένη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε πολύ σημαντική μείωση στον αριθμό ε, και του χρόνου και των καταβολών που απαιτούνται στην εμπορική δραστηριότητα. Αυτό που είδαμε λοιπόν ότι καθώς οι χώρες βελτίωσαν τις φορολογικές τους υπηρεσίες παντού, πέρασαν κάποιε από τα ωφελήματα και στην επιχειρηματική κοινότητα μειώνοντα κάποιου φορολογικού συντελεστές. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην υποσαχάρια Αφρική, όπου σε πολλέ χώρε ήταν παράλογα υψηλή συντελεστή φορολογία, τόσο υψηλή που κανεί δεν πλήρωνε ουσιαστικά. Υπήρχαν κάθε είδου τρευλώσει τη αγορά και όλοι περνούσαν σε ε, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Καθώ βελτιώθηκε λοιπόν οι φορολογικέ ε, διοικησει, βελτιώθηκε κατά πολύ, ε, μειώθηκαν οι οι φορολογικοί συντελεστέ ε, πολύ ισχυρά σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Και εν κατακλείδη σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, εδώ ένας ε, δείκτη σε ό,τι αφορά την καταγραφή ε, ιδιοκτησίας, υπήρξε μείωση ε, του χρόνου που απαιτείται για την καταγραφή ε, ιδιοκτησία σε όλο τον πλανήτη. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί και πάλι οι εμπειρικέ μελέτε δείχνουν ότι χώρε που έχουν πολύ καλά καθεστώτα πνευματική ιδιοκτησία είναι ακριβώ χώρε που θα επενδύσουν περισσότερο επιχειρήσει, όπου η επιχειρηματική κοινότητα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία για εχέγγυα, επομένω τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων στι χώρε αυτέ και αντίστοιχη μόχλευση, αν θέλετε, τη οικονομία. είναι όλες αυτές τις φορές του Μανώντο Ντεσότο που έγραψε ένα βιβλίο πριν από κάποια χρόνια με τίτλο «Το μυστήριο του κεφαλαίου» που ακριβώς ε, κατέδειξε πόσο σημαντικά είναι τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εξασφάλισης είναι σημαντικά γιατί έχουν πραγματικές μακροοικονομικές ωφέλειες. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την ε, ε, εξέλιξη του σχετικού δίκτυ στη μελέτη αυτή. Εάν με, μία με ένα λόγο θα ήθελα να συνοψίσω τις 300 ε, σελίδες της έκθεσης αυτής, θα ήταν η λέξη σύγκληση. Είναι ίσως η πιο σημαντική χάρτα αυτή της παρουσίασής μου εδώ. Θα ήθελα εντάχει να σας επισημάνω αυτά βλέπετε στο γράφημα στην πάνω αριστερά αγωνία, αν και ισχύει εξίσου και για όλες τις άλλα γραφήματα τρία γραφήματα και δεν ξέρω ποια άλλα γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι ότι πήγαμε στο δείγμα του 2005 και το χωρίσαμε σε δύο ομάδες. Το χειρότερο ε, 25% τις χώρες δηλαδή όπου η χρηματική νομοθεσία είναι η πιο βαριά και πολλές φορές η πιο, η πιο πολύπλοκη και ακατανόητη και αποκλείσαμε αυτό το, το κάτω 25% και το άνω 25%. Κρατήσαμε λοιπόν το χρόνο, ε, το δείγμα, με το χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Στο χειρότερο ήταν 105 μέρες, ενώ στο καλύτερο ταρτιμόριο ήταν 29 μέρες. Τις επόμενα χρόνια βλέπουμε μια, ε, ένα κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ αυτών των ομάδων χωρών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπουμε μια διαδικασία το 2012 το, η ψαλίδα αυτή έκλεισε πάρα πολύ. Εξακολουθεί να είναι μεγάλη, αλλά πολύ μικρότερη από αυτό που ήταν το 2005. Και περί αυτού πρόκειται στη μελέτη αυτή το επιχείρημα 2012. Ή δηλαδή να ενθαρρυνθούν οι χώρες που είναι στο χειρότερο ταρτιμόριο, όπου οι διαδικασίες είναι οι πλέον δύσκολες, οι πλέον επαχθείς, οι πλέον πολύπλοκες, που εισάγουν και τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην αγορά, τι ενθαρρύνουν να εισάγουν κάποιες από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές στις χώρες όπου βλέπουμε που έχουν το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σύγκλησης το βλέπετε σε όλους τους δείκτες, σε όλο τον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το project αυτό, το επιχειρήν, ε, υπήρξε τόσο επιτυχές στην προώθηση μεταρρυθμίσεων. Και, το, και περιμένουν την έκθεση αυτή κάθε χρόνο όλοι οι πολιτικοί θύνοντες ανά τον κόσμο. Αυτό είναι ένα γράφημα στο οποίο έχουμε συμπεριλάβει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν παρουσιάζουμε μόνο το χειρότερο και το βέλτιστο ε, τεταρτημόριο σε ό,τι αφορά τον δίκτυο αυτό, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπάρχει βελτίωση στο μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια προσεγγίζει περισσότερο το βέλτιστο τεταρτημόριο από ότι το ε, χειρότερο και σε ορισμένε περιπτώσει ε, ανήκει και στην ομάδα. Κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν στο βέλτιστο αυτό αρθμόριο. Κοιτάω το ρολόι γιατί θέλω να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε και χρόνο για συζήτηση. Μια από τι προκλήσει. Ναι, αν θέλετε λίγο όμω, δεν χρειάζεται να βιαστείτε, γιατί έχουμε, έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση, οπότε μην, δεν χρειάζεται να πιέζεστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στην Παγκόσμια Τράπεζα είναι ότι στο project αυτό ε, βαθμολογούμε τις χώρες. Δηλαδή, στο συνοπτική περίληψη της έκθεσης αυτής υπάρχει ο πίνακας 1-1 που παρουσιάζει μια βαθμονόμηση όλων των χωρών. Αναφέρουμε ποια είναι 1, 2, 3, 10, 185, 195 φέτος. Ε, αυτός ο πίνακας είναι λίγο αντιφατικός, δηλαδή έρχονται αξιωματούχοι στην Παγκόσμια Τράπεζα και λένε, όπως μου είπε για μένα η Ινδονησία για παράδειγμα φέτος το Ιανουάριο, ότι κοιτάξτε έχουμε εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει το άλλο και έχει πραγματικά αλλάξει πάρα πολύ η βαθμολογία μας και μπορεί να αποθαρρυνθούν τελικά από την έκδοση του τελικού πίνακα. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι πίνακε αυτοί είναι σχετικοί από τη φύση του. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να προοδεύει, αλλά αν υπερπατά δηλαδή ουσιαστικά και άλλε χώρε στην περιοχή σου τρέχουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο, παραμένει πάλι πίσω. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να σημειώνει πρόοδο, αλλά παρόλα αυτά να παραμένει πίσω. Πέρσι λοιπόν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ω ομάδα αν υπάρχει ένα άλλο τρόπο να παρουσιάζουμε τα στοιχεία πέραν τη βαθμολογία αυτή που να μπορεί να δίνει μια διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά την πραγματική επίδοση των χωρών αυτών σε σχέση με τους δείκτες. Κάναμε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα άσκηση και θέλω για λίγο να σας το παρουσιάσω αυτή, γιατί θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο αυτού την ανάλυση στην έκθεση αυτή και γιατί επίσης ε, είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη η ανάλυση αυτή. Δηλαδή οι κρατικές αρχές, οι υπουργοί δεν υπερβάλλουν, πραγματικά σωσμένες φορές εξέφρασαν ενθουσιασμό για αυτές τις ε, μήτρες. Ε, μπορεί να φαίνεται λίγο εκφοβιστικός ο πίνακας αυτός, αλλά προσέξτε τον παρακαλώ πολύ, θα δείτε ότι ε, κατά βάση είναι μια πολύ απλή ιδέα. Επειδή πέρσι είχαμε στοιχεία 9 ετών για 180 σχεδόν χώρε, αρχίσαμε να ρωτηθούμε, να αναρωτιόμαστε πού μπορούμε να βρούμε τι καλύτερε επιχειρηματικέ πρακτικέ. Για παράδειγμα, έχουμε έναν δείκτη που έχει τίτλο δικτυ που εχει τιτλο εφαρμογη ε, των συμβάσεων» είσαι επιχειρηματίας, έχει πρόβλημα με κάποιο προμηθευτή, καταβάλει χρήματα, Αυτό ουσιαστικά δεν σου αποστέλει τα, τα προϊόντα τα οποία έχει υποσχεθεί, θέλεις και καταφεύγεις δικαστικά. Πόσο χρειάζεται, πόσο χρόνος χρειάζεται για να εφαρμοστεί πραγματικά μια εμπορική συμφωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια επιχειρηματική κοινότητα. Για την Σιγκαπούρη χρειάζονται 150 μέρε. Είναι ο βέλτιστο και μικρότερος χρόνο. Υπάρχουν χώρε, συμπεριλαμβανομένων και χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρειάζονται χρόνια για να επιληθεί και πραγματικά να εφαρμοστεί μια εμπορική συμφωνία. Η χρονική λοιπόν συνιστόσα, η Σιγκαπούρα μα δίνει την καλύτερη πρακτική. Μετά αναρωτηθήκαμε, υπάρχουν χώρε όπου δεν στοιχίζει τίποτα για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Ναι, στη Δανία και τη Σλοβενία, εάν θε να ξεκινήσει μια επιχείρηση, σου στοιχίζει ακριβώ μηδέν. Στη Νέα Ζηλανδία χρειάζονται, απαιτούνται λίγα δολάρια, αν και στη Ζηλανδία χρειάζονται μόνο μία μέρα και μία διαδικασία. Δηλαδή με το που κλικάρεις, ε, χτυπάς την ε, online πλατφόρμα, αμέσως θα σε χρεώσουν μια απειροελάχιστη αμοιβή που καλύπτει τα κόστη ε, διαχείριση του συστήματος. Βλέπουμε δηλαδή, αυτό ισχύει και για τους 40 δείκτες που έχουμε στην έκθεση αυτή. Και τελικά φτάνουμε αυτή την έννοια που την ονομάζουμε το όριο. Είναι αυτή η γραμμή που κινείται από αριστερά προς τα διάξια, από 0 έως το 100. Είναι μια υβριδική μήτρα, αν θέλετε, η οποία βασίζεται στο δείγμα, σε πραγματικούς αριθμούς που προέρχονται από δειγματοληψία από στοιχεία 9 ετών. Αφήστε τη το κάνεις αυτός, μπορείς πάλι να ανατρέξεις το 2005 και να πεις πόσο απέχει μια χώρα από το όριο. Αυτές είναι οι μικρές ε, μπλε κουκίδες που είναι στο χαμηλότερο όριο και κάτω από τη γραμμή αυτή που κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Και το επόμενο ερώτημα που μπορεί να θέσει είναι ότι εάν φτάσει το 2012, πόσο έχει μειώσει την απόστασή της μια χώρα από το όριο. Και αυτές είναι οι μικρές ακίδες που βλέπετε πώς οι χώρες δηλαδή κινήθηκαν προς την κατεύθυνση μίκνησης ε, της απόστασής τους από το όριο αυτό. Αυτό που θα παρουσιάσουμε στο γράφημα αυτό είναι ότι οι περισσότερες χώρες, με εξαίρεση χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Ζιμπάμπουα, Ζιμπάμπουε που είχαν επιδείνωση του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος το 2012 από το 2005, οι περισσότερες άλλες χώρες σημείωσαν πρόοδο, μικρή ή μεγάλη. Και αυτό είναι ουσιαστικά ο λόγο για τον οποίο στι χώρε αρέσει ιδιαίτερα ο πίνακα αυτό αυτή η μήτρα. Γιατί λένε, α ξεχάσουμε του ίδιου, α ξεχάσουμε την Νέα Ζηλανδία, α ξεχάσουμε την ιδέα τη Σιγκαπούρα. Εάν είσαι ένα αξιωματούχο στην υποσαχάρη Αφρική, δεν έχει κανένα νόημα να σου λένε κάθε χρόνο ότι η Σουηδία έχει καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον από σένα, από τη δική σου χώρα. Αυτό το ξέρει. Σε βοηθά όμω ιδιαίτερα να, να αποτιμάται και να βλέπει πραγματικά ότι τώρα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από το 2005. Αυτό είναι αθαρρυντικό, γιατί κατά σου λέει ποια είναι η επίδοσή σου σε σχέση με το δικό σου ιστορικό. Ποια είναι, δηλαδή, ποιοι είναι οι καρποί τη προσπάθειά σου. Φέτος λοιπόν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε και να ε, δημοσιεύσουμε αυτό το πίνακα στην έκθεση που είναι εκπληκτικά επιτυχημένος. Λέει δηλαδή ότι αυτές είναι οι 50 χώρες που είχαν την μεγαλύτερη ε, σμίκρινση της ε, απόστασης. Πού είναι η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, πουθενά. Γιατί, Γιατί είχαν ήδη καταπληκτικό επιχειρηματικό περίμα 2005, ως εκ τούτου μείωσαν μεν λίγο την απόστασή τους από το όριο, όχι πολύ, λίγο, αλλά είχαν λίγο περιθώριο. Ενώ χώρες όπως η Γεωργία, η Ρουάντα και, πάρα, και χώρε όπω Αφρική σημείωσαν τεράστια πρόοδο και αναφέρονται στον πίνακα αυτό λόγω ακριβώ τη προόδου που σημείωσαν σε σχέση με το ιστορικό του. Όλο και περισσότερο λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή την ανάλυση στην έκθεση του επιχειρήν, γιατί του αρέσει ο πίνακα αυτό και είναι πιο ενθαρρυντικό. Να σας δείξω τώρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα του είδους της ανάλυσης που κάποιος μπορεί να έχει με, την, ε, με τον πίνακα αυτής τη μήτρας και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτόν τον πίνακα γιατί έχει ενδιαφέρουσα ιστορία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε τις 7 ε, περιοχές του κόσμου που χρησιμοποιούμε ε, για την ταξινόμηση των χωρών και πάνω πάνω βλέπετε τον ΩΣΑ. Είναι η περιοχή που έχει τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές στον κόσμο. Είναι η περιοχή που είναι πιο κοντά στο όριο. Βελτιώθηκαν από το 2005 στο 2012. Τώρα, θέλω όμως να εστιάσετε στην ε, γραμμή με τις μαύρες κουκίδες από αριστερά προς τα δεξιά, ήταν στην τέταρτη γραμμή του 2005, κεντρική και ανατολική Ασία και έχει ανέβει στη δεύτερη θέση το 2012. Είναι μια περιοχή η οποία πλησίασε, ήταν η περιοχή που πλησίασε πιο γρήγορα το όριο. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε, το, ο πίνακας αυτός είναι ε, πολύ εύγλωτος, αλλά αναζητήσαμε τι συνέβη. Ε, δύο πράγματα συνέβησαν σε αυτή την περιοχή. Ε, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και την κεντρική Ασία. Και κυρίως αφορά τις χώρες κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει είναι δύο πράγματα. Έχουμε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία, Λετωνία, Λιθουανία, ε, χώρες οι οποίες μπήκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησαν σημαντικές ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί, γιατί αυτό ήταν το τίμημα για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ξεκίνησαν, ε, δημιούργησαν καλές μεταρρυθμιστικές συνήθειες, να το πούμε έτσι, και συνέχισαν με μικρές διαφοροποίησεις μεταξύ των χωρών. Για αυτές οι χώρες για διαφορετικούς λόγους πλέον, γιατί για παράδειγμα πρέπει να ανταγωνιστούν τη Γερμανία, τη Σουηδία κλπ. Ε, συνεχίζουν τις μεταρρυθμίσεις ανεξαρτήτως από την ανάγκη εισόδου πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συνεχίσει λοιπόν αυτό το μονοπάτι. Και φέτος μάλιστα η Πολωνία μεταξύ των 185 χωρών που καλύπτουμε ήταν η χώρα που πιο πολύ κάλυψε απόσταση μέχρι το όριο. Αυτό αναζητούμε πάντοτε αυτή τη χώρα κάθε χρόνο. Φέτος ήταν η Πολωνία. Μετά έχουμε Κροατία, Μακεδονία, λέει Σερβία, Μαυροβούνιο. Μια δεύτερη ομάδα χωρών που θα είναι μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσει ενταξιακέ ή προενταξιακέ, και κάνουν αυτό που έκαναν οι χώρε τη Κεντρικής και Ευρώπης πριν από μια δεκαετία. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή, ορισμένε χώρε πιο γρήγορα από κάποιε άλλε, αλλά η κατεύθυνση τη αλλαγή είναι σαφή. Μεταξύ αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι μεταρρυθμίσεις που πραγματικά έχουν σχέση με τους δείκτε που χρησιμοποιούμε. Αν τα δείτε όλα αυτά μαζί, θα καταλάβετε την σύγκληση της κεντρικής και Ανατολική Ευρώπη προ τι καλέ, βέλτιστες επιχειρηματικέ πρακτικέ. Και αυτός ο πίνακας προέρχεται από την έκθεση και θέλω να σας τον ε, υπογραμμίσω γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, η, ε, ε, η μάρκα Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πληγεί κατά κάποιο τρόπο για λόγους δημοσιονομικών προβλημάτων κλπ. Και αυτός ο πίνακας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πείραμα που βοηθάει τις χώρες να βελτιωθούν. Αν δείτε τις χώρες που τα τελευταία 50 χρόνια πέρασαν από χαμηλό εισόδημα σε υψηλό επίπεδο, είναι γύρω στι 25 χώρες, οι μισές από αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτός ο πίνακα μα υπενθυμίζει μέσα στη σκοτεινιά και το ζόφο που ζούμε, σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι μια πολύ καλή μηχανή σύγκλησης. Αυτό δεν το βλέπουμε στην υποσαχάρη Αφρική για παράδειγμα. Είδατε το βιβλίο του καθηγητή Collier, ε, το κάτω ένα εκατομμύριο είναι ο τίτλος, ε, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Κοιτάει τις 58 χώρες που βρίσκονται πιο χαμηλά, ε, με πληθυσμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο άτομα. Ε, και αντί να συγκλίνουν, αποκλίνουν. Αποκλίνουν από το μέσο όρο του υπόλοιπου κόσμου. Κάτι που δημιουργεί διάφορα προβλήματα για τη διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ πιο επιτυχές παράδειγμα σύγκρισης. Θέλω να τελειώσω δείχνοντας σας ένα ακόμα πίνακα. Δεν είναι ακριβώς ένας πίνακας, θα σας πω και ίσως ε, μετά την, μετά, αφού σας πω την ιστορία πίσω από τον πίνακα θα σα πω και κάτι πιο προκλητικό. Το 2009 ε, τα μέλη του, της Συνασίας Ασίας και Ειρηνικού, 29 χώρες, ε, αποφάσισαν να κάνουν το επιχειρήν πιο γρήγορο ή πιο φτηνό κατά 25% μέχρι το 2015 με δείκτες επιχειρηματικότητα που θα του βοηθούσαν να ποσοτικοποιήσουν τα πράγματα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, έχουν πετύχει του στόχου του μέχρι τώρα. Έχουν ομάδε εργασία που συναντώνται δύο φορέ το χρόνο. Μερικέ φορέ συναντιόμαστε μαζί του και του δίνουμε τεχνική συνδρομή. Θα πετύχουν το στόχο του για το 2015 αν συνεχίσουν αυτό που έχουν κάνει τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, τι, τα επόμενα τρία χρόνια. Ε, όταν πήγα στην Ινδονησία, ο Υπουργός Οικονομικών μου είπε ότι το 2009 η περιοχή αυτή είχε επιλέξει έξι πρωταθλητές. Ιαπωνία, Καναδάς, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες. Τους, αυτούς τους καλύτερους επιχειρηματικούς προορισμούς. Και αυτές οι έξι χώρες είχαν αποφασίσει να παράσχουν τεχνική συνδρομή στις υπόλοιπες χώρες του τόξου του ειρηνικού. Στην Ινδονησία λοιπόν ο υπουργός μου είπε οι Κορεάτες μας παρέχουν ε, τεχνική συνδρομή για την εκτέλεση συμβολέων. Η Κορέα έχει ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα, δικαστικό σύστημα, σύστημα επίλυση διαφορών κλπ. από ότι εμείς. Και από τη μια μεριά ευγνωμονούσε τους Κορεάτες και από την άλλη μεριά λίγο φοβισμένος διότι οι Κορεάτες έλεγε είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί, ε, απαιτητική. Πάντως η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας από τη μία χώρα στην άλλη μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης και αδελφότητας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και εξετάσαμε ε, την κατάσταση πιο βαθιά και τις πληροφορίες περιλάβαμε. Ε, η Ιαπωνία έχει δώσει συνδρομή στην Ταϊλάνδη ας πούμε. Ο Καναδάς ε, σε ορισμένες άλλες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν διμερείς ε, εταιρικές σχέσεις που προέκυψαν από αυτή την προσπάθεια. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα, σε ένα περιβάλλον πολύ θερμό. Και όλα αυτά ε, εκτός Παγκόσμιας Τράπεζας. Ε, Εμεί δεν κάναμε τίποτα. Μαζέψαμε τα στοιχεία, τα ανεβάσαμε στο site μας, τα βάλαμε στις εκθέσεις μας. Άλλες χώρες τα χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, ε, αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα. Και βλέπετε πώς επηρέασε το project μας στον κόσμο. Τέλος, να, σας, ε, να μοιραστώ μαζί σας και αυτή την ιδέα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο, να λάβει μια παρόμοια πρωτοβουλία. Αφού το κάνει η ΑΠΕΚ, δηλαδή οι χώρες του ε, τόξου του ειρηνικού, που δεν έχουν μια περίπλοκη ε, ε, δομή ε, οργάνων, θεσμικών οργάνων, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένων των προκλήσεων ανταγωνιστικότητα που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Ξέρετε ότι πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υψηλό χρέο. Πώ θα βγουν από αυτήν την κατάσταση, θα βγουν μέσω τη ανάπτυξη και αυτή θα είναι η μηχανή αντιμετώπιση του προβλήματο ε, του χρέου. Πρέπει το ΑΕΠ να αυξηθεί έτσι ώστε να μειωθεί ο λόγο χρέου προ το ΑΕΠ. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, στι ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ε, και οι δύο αυτές χώρες είχαν ε, χρέος ε, παραπάνω από το 100% του ΑΕΠ τους με την ανάπτυξη έλυσαν το πρόβλημα αυτό, αυτή θα είναι η λύση και για την Ευρώπη. Και αυτό δεν θα γίνει αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν γίνουν πιο ανταγωνιστικές, δεν δημιουργήσουν πιο φιλικό προς, τις, ε, προς το επιχειρήν περιβάλλον. Μόνο έτσι θα αυξηθεί και η απασχόληση. Δεν πρόκειται να γίνει αν δεν αντιμετωπιστούν κάποια από τα θεμελιώδη προβλήματα, θεμελιώδης περιορισμούς που υφίστανται αυτή τη στιγμή και ε, τα οποία μετράει το project επιχειρήν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έτσι ολοκλήρωσα την ομιλία μου. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την έξοχη παρουσίαση και πολύ εμπεριστατωμένη για τις ε, εξελίξεις του προγράμματος Επιχειρήν 2013. Το παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η Κριστιανά Μοσκαρντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά γιατί η έκθεση πραγματικά ήταν εξαιρετικά αναλυτική. Πιστεύω ότι απεικονίζει την έρευνα την οποία κάνατε, όπου επί τη βάση αυτής θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις σε ό,τι μας αφορά. Γιατί όπως Γιατί υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης στο 2. Μέχρι ότου, βρω το αγγλικό κανάλι, νομίζω ότι είχα το ολοκληρώσει. Μήπως θα μπορούσατε να επαναλάβετε. Θα μπορούσατε να επαναλάβετε. Ναι, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ σημαντική και ε, ενδελεχέστατη έκθεση που μας παρουσιάσατε και για την οποία πιστεύω ότι πρέπει, επί τη βάση της οποίας θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να λάβουμε κάποιες αποφάσεις επί τη βάση των στοιχείων που από τη μία μεν μπορούν να είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, αλλά από την άλλη μπορούν να είναι και ανησυχητικά. Δεδομένου ότι από την έρευνα ε, συνάγουμε ότι εκεί όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος, περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, πολύ περισσότερα χρήματα για να συσταθεί μια νέα επιχείρηση, εκεί ακριβώς που συμβαίνουν όλα αυτά υπάρχει και περισσότερη διαφορά. αυτό μας δίνει ένα νέο στοιχείο και σε ό,τι αφορά τις ε, διμερείς μας συμφωνίες, ώστε, ως μέτρο δηλαδή αξιολόγησης των συμφωνιών αυτών. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση συμφωνιών που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, υποστηρίξαμε ότι προτού συναυθεί κάποια συμφωνία, διμερή συμφωνία, θα πρέπει να αξιολογήσουμε διάφορες πτυχές από το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων μέχρι την αξιοπιστία του εταίρου. Σήμερα όμως με την έκθεση που μας παρουσιάσατε, με την έρευνα αυτή την οποία μας παρουσιάσατε, έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία και παραμέτρους πάνω στους οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Εάν μια χώρα έχει μια πολιτική τάξη στην ε, η οποία η διαφθορά μπορεί να είναι μετρήσιμη ακόμα και μέσω του γραφειοκρατικών επιπλοκών και της χρονοτριβής που ε, υπάρχει και που απαιτείται σε μια χώρα για να συσταθεί μια νέα επιχείρηση ή συναρτήσει του κόστους που ε, συνεπάγεται, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και μέτρο ακριβώς ε, εξέτασης ε, κάποιας συμφωνίας, όταν δηλαδή θα κάνουμε τις ε, σχετικές μας αξιολογήσεις για τις προσεχείς διμερείς συμφωνίες. Δεύτερο σημείο, η χρόνη καταβολών. Αυτό με κάνει να σκεφτώ και την δική μας ευρωπαϊκή απόφαση να ζητήσουμε από την Ευρώπη χρόνους ε, πληρωμών μέσα στο 30ημερο. Δεν ξέρω τι αποτιμήσετε στους διάφορους τιμής, τομείς, αλλά μπορώ να πω ότι σε ό,τι αφορά τον γεωργικό τομέα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, ήδη έχουν δημιουργηθεί καρτέλ των πιο σημαντικών επιχειρήσεων ε, διανομής, των πολύ μεγάλων δηλαδή ε, εταιριών ε, διανομής, για τους οποίους τα 30 μέρες δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή στους γεωργούς, αντί να πληρώσουν εγκαίρος, είτε πληρώνουν πάρα πολύ αργά, είτε τους επιβάλλουν προκειμένου να πληρώσουν μέσα στο 30 μέρες, αντί να πληρώσουν ένα ευρώ, τους πληρώνουν ένα κλάσμα του ένα ευρώ, διαφορετικά θα επιλέξουν άλλο προμηθευτή. Και νομίζω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες συγκεκριμένε δράσεις ελέγχου, που είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, είναι δυνατόν να μας πείτε σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία ή σε σχέση με ασιατικές χώρες, τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, έχουμε συμφωνίες, μπορείτε να δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία από αυτά που μας δώσατε. Φρανσέσκα Ευχαριστώ. Δεν είμαι πρώτη πιστεύω που θίγω αυτό το ζήτημα. Εσείς μας παρουσιάσετε μια έκθεση για ορισμένου δείκτες, ε, εάν γίνονται σεβαστοί, δεν γίνονται, αν εφαρμόζονται ή όχι, ειδικοί μετρήσιμοι δείκτες που εφαρμόζονται ε, για τη μελέτη κλπ. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα πίσω από τα διάφορα αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία. Ας πούμε, ε, η νομιμότητα ετοιμάτων, οι καθυστερήσεις καταχώρησης νέων επιχειρήσεων, ε, διαβουλεύσεις ή συζητήσεις που πρέπει να γίνουν συμβουλευτικής φύσεως που δεν είναι κάτι κακό και υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις ε, στη ε, διανομή των κονδυλίων υπάρχουν καθυστερήσεις σε εμά, αλλά εμεί κάνουμε και ενδελεχείς ελέγχους επειδή έχουμε έλεγχο από τους φορολογούμενους και έχουμε και την κοινοβουλευτική διαδικασία που μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει ότι τα πράγματα θα συζητηθούν πολύ λεπτομερώς. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν όλα αυτά τα ζητήματα παίζουν κάποιο ρόλο στην έκθεσή σας, εκτός από όλα τα μετρήσιμα στοιχεία για το πόσες μέρες χρειάζεται για να εδραιωθεί μια νέα επιχείρηση, για την εκτέλεση συμβάσεων κλπ. κλπ. Λαμβάνετε ε, ε, υπόψη και αυτά τα παράπλευρα ζητήματα στη μελέτη σας. Ευχαριστώ, Πίτερ Στάσνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς ε, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την παρουσίαση και τον αριθμό των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάσατε. Ε, το ερώτημα μου είναι, εάν οι στατιστικές συνδέουν άμεσα τις επιχειρήσεις το επιχειρησιακό περιβάλλον και τη βελτίωσή του με την βελτίωση των στοιχείων του ΟΕΠ κάτι δηλαδή το οποίο μπορείτε εσείς να προσφέρετε στις χώρες αυτές ε, ως συμβουλή ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κάτι το εφαρμόσιμο. Και δεύτερον, μπορείτε να βοηθήσετε, να συστήσετε σε αυτούς που είναι στο, στον πάτο των πινάκων ή των κατατάξεων πώς μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο με την προσέγγιση των χωρών του APEC, Ασίας Ειρηνικού, ε, προτιμάτε μια προσέγγιση διμερής ή ε, συμμετέχετε άμεσα στην παροχή συμβουλών ε, προς τις χώρες αυτές και βοήθειας. Ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ορισμένα ερωτήματα σε εσάς. Ε, λόγω πίεσης χρόνου νομίζω δεν παρουσιάσατε μία από τις διαφάνειες για τις νότιο ε, ευρωπαϊκές χώρες, τις μεσογειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης που ε, έχουν κατά κάποιο τρόπο εκτεθεί, εκτεθεί και ντροπιαστεί. Είναι, είναι μία από τη διαφάνεια που βλέπω εδώ στις συνομιλίες σας που δεν είδαμε. Το θέμα είναι πώς μπορούν να σπρώξουμε τις χώρες αυτές να προσπαθήσουν πιο δυνατά, πιο πολύ, διότι το ε, χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτών και των υπόλοιπων χωρών ε, μειώνεται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Σε μία χώρα σε μια χώρα μειώνεται το χάσμα αυτό και αυτό είναι πολύ καλή θετική είδηση υπό το μακροοικονομικό, μακροπρόθεσμο οικονομικό πλαίσιο. Μία από τις χώρες αυτές λοιπόν μειώνει το, το, το, το χάσμα, το κενό, τις διαφορές που υπάρχουν με τις άλλες χώρες. Τι άλλο μπορεί να γίνει λοιπόν. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι πιο προκλητική. Από ό,τι κατάλαβα, το μήνυμά σας είναι το εξής. Λιγότεροι ε, κανονισμοί, τόσο όσο, λιγότερο, όσο μικρότερο είναι το κανονιστικό πλαίσιο, τόσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί να είσαι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορείτε να απευθύνετε στις κυβερνήσεις όλων των ε, χωρών ε, στον κόσμο. παραδείγματος χάρη ε, λιγότερο κανονιστικό πλαίσιο στο φορολογικό, στο οικονομικό, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των χωρών παγκοσμίω. Και με αυτό την πρόκληση ολοκληρώνω. Και σας δίνω και πάλι το λόγο. Um, ευχαριστώ πολύ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα τις απαντήσω με κάπως διαφορετική σειρά. Θα αρχίσω με ε, το ερώτημα που τέθηκε για τη Νότια Ευρώπη. Ναι, βεβαίως, νοτιοευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και βελτιώνονται και τις παρακολουθούμε τις βελτιώσεις αυτές και έχουν συμπεριληφθεί στις, στην προσέγγιση μας την τελευταία έξεση. Ιδιαίτερα αναφέρουμε στην Ιταλία και στην Ελλάδα που έχουν βελτιώσει την κατάταξή τους σημαντικά. Από 100η θέση στην 78η είναι σήμερα Ελλάδα, από 87η είναι τώρα 73η η Ιταλία. Αυτές είναι πολύ σημαντικές βελτιώσεις και αυτό βασικά αντανακλά την αναγνώριση και κατανόηση από πλευρά των αρχών στις χώρες αυτές ότι πρέπει να δημιουργήσουν ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα, ότι πρέπει να διευκολύνουν το επιχειρήν και ότι πρέπει να απαλλαγούν από πάρα πολλά ε, προσκόμματα λόγω ενός κανονιστικού υπερφορτωμένου πλαισίου. Έχω πει και στις δύο χώρες. Και στη Ρώμη και στην Αθήνα συναντήθηκα με, υπουργούς, με υπουργούς και στις δύο χώρες και με ενθαρρύνει ιδιαίτερα η προσέγγιση τους. Δηλαδή αναγνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία έχουν στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και του κανονιστικού, των κανονιστικών προσκομμάτων και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι αυτά τα, τις εξελίξεις τις κρίνουμε εμείς ως αρνητικές, αλλά πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να διατηρηθούν για πολλά χρόνια. Οι χώρες που έχουν πραγματικά προχωρήσει, έχουν κάνει βήματα στο επιχειρήν, στη διευκόλυνση κλπ. Χρειάζονται τρία με πέντε χρόνια για, την, ε, για τις μεταρρυθμίσεις τους να μπορούν να είναι μετρήσιμες. Δηλαδή για να δούμε τα αποτελέσματα δεν γίνεται αυτό σε μια νύχτα. Παραδείγματο χάρη, όλοι οι κανονισμοί για περιχρεοκοπία, ε, για τις επιχειρήσεις κλπ. Όλα αυτά αποτούν μια μακροχρόνια προσέγγιση, όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και πάρα πολλές τεχνικές διοικητικέ προσαρμογές για να μπορέσουν και τα δικαστήρια να ανταποκριθούν στις ε, νέες ανάγκες της ε, παρακολούθησης ε, των προσφυγών, εκτέλεσης συμβάσεων κλπ. Εφαρμογής όλων αυτών των κανονισμών. Και το μέλος που ο πρόεδρος που ανέφερε αυτό το, το ερώτημα είχε πάρα πολύ δίκιο, δεν το ανέφερε. Αυτή τη διαφάνεια δεν την ε, ε, έδειξα για να μην μακρηγορήσω περαιτέρω. Τώρα, ε, εάν εμείς προσφέρουμε συμβουλές και τεχνική βοήθεια σε χώρες οι οποίες χρειάζονται βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος ή εάν αυτό επαφίεται σε ίδιες πρωτοβουλίες όπως το πλαίσιο του ΑΕΠΕ, Κασίας Ειρηνικού, έχουμε μια συμβουλευτική η υπηρεσία δεν ε, την εκτελώ, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Εμείς κάνουμε ε, εκθέσεις, ε, κάνουμε την έρευνα, στοιχεία, διατυπώνουμε, συντάσσουμε τις εκθέσεις. Αλλά υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη διεύθυνση και ο Πιέρ Γκισλάν είναι διευθυντής αυτής της μονάδας, είναι και μάλιστα, ο οποίος διευθύνει αυτή την συμβουλευτική ομάδα και πηγαίνει σε χώρες οι οποίες λαμβάνουν πολλές φορές και επιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και οι δείκτες μας δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση τεχνικής βοήθειας και η Παγκόσμια Τράπεζα το κάνει αυτό, αλλά υπάρχει ένα συνικό τείχος μεταξύ της δικής μου διεύθυνσης και της διεύθυνση του Πιέρ, διότι εμείς κάνουμε τη συλλογή και ανάλυση ε, στοιχείων και τα οποία παραδίδουμε μέσω εξέσεων μετά στην παγκόσμια κοινότητα και ο Πιέρ κάνει τη συμβουλευτική δράση. Ε, το, μάλιστα αυτή η διεύθυνση η παροχή συμβουλών και βοήθειας και λοιπά είναι μεγαλύτερη σε προσωπικό γενικά είναι μεγαλύτερη από τη δική μου για να σας δώσω δηλαδή μια εικόνα των διαστάσεων. Μία άλλη ερώτηση αφορούσε πώς η βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να παρακολουθηθεί από τη βελτίωση των δικτών ε, για την προσαρμογή των δικτών. Ναι, βεβαίως, έχουμε αρχίσει, έχουμε ξεκινήσει να παρακολουθούμε τους δίκτες ανάπτυξης και στη φετινή έκθεση έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Εξετάζοντας εάν το επιχειρήν και η κατάταξη βάσει του επιχειρήν συσχετίζονται με τον όγκο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Και ε, διαπιστώσαμε ότι ο συσχετισμός αυτός είναι τόσο υψηλός, ώστε αξίζει τον κόπο να δημοσιεύσουμε μία μελέτη περιπτώσεων που μπορείτε να έχετε. Όσο προχωρούμε προς τα πάνω στην κατάταξη του επιχειρήν, βλέπουμε ότι τόσο βελτιώνεται και η κατάσταση ροών ξένων άμεσων επενδύσεων, επενδύσεων κατά κεφαλή. Πράγματι υπάρχει λοιπόν αυτό το συσχετισμός και οι δείκτες που χρησιμοποίησαμε για να μετρήσουμε αυτές τις δύο, αυτά τα δύο βήματα, αν θέλετε, αυτές τις δύο στήλες είναι οι δείκτες ακριβώς του, της μεθόδου Frontier. Οι χώρες οι οποίες έχουν μειώσει τη διαφορά αυτή ε, του συσχετισμού δείχνουν ακριβώς ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ έχει προχωρήσει ταχύτερα και τα, όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα ε, τα οποία είναι τεχνική φύση θα δημοσιευτούν του χρόνου. Ε, έχουμε, συλλέγουμε σε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι ότι έχουμε τον κατάλληλο τρόπο να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτά φέτος, άρα θα γίνει αυτό του χρόνου. Και μια άλλη ερώτηση για το αν ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα έχει, είναι προκατηλημένο, είναι αντικανονιστικό, αντιρυθμιστικό και αν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε τα ε, ρυθμιστικά πλαίσια σε όλες τις χώρες. Όχι βέβαια είναι η απάντηση. Αν δούμε τις χώρες που ε, έχουν το καλύτερο επιχειρήν, το καλύτερο περιβάλλον, τότε θα δείτε ότι δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν απελευθερώσει τα πάντα, ε, εις βάρος της ασφάλειας, εις βάρος ε, του, του, του ασφαλούς περιβάλλοντος, εις βάρος ε, των ευθυνών που έχουν ενάντια της κοινωνίας των πολιτών. Όχι. Απλώς έχουν εφαρμόσει την έξυπνη ε, τους έξυπνους κανονισμούς, τους, το, το έξυπνο ρυθμιστικό πλαίσιο με έναν τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί λογικός. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε ένα κάπως αφηρημένο περιβάλλον. Ας πούμε για τις άδειες κατασκευής. ή χώρες οι οποίες έχουν ένα πολύ καλό καθεστώς για την ε, άδεια στις ε, πολλοδεμή, την άδεια οικοδομών, οικοδομών κατασκευής κλπ. Χρησιμοποιούν, λειτουργούν σαν μία μικρή αποθήκη. Παραδείγματο χάρη, άμα ένα οξύ μία μικρή αποθήκη, δεν έχεις μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. εάν ομω χτιζει ένα μία μεγάλη βιομηχανία, ένα εργοστάσιο, που θα ασχολείται με, την, ε, χημικά απόβλητα, αναπόθεση ή το οποίο θα, έχει, θα ρηπαίνει το περιβάλλον, χρειάζεται βεβαίως ένα πολύ πιο αυστηρό ε, πλαίσιο παροχής αδειών ε, κατασκευής. Άρα λοιπόν όλο αυτό το καθεστώς της παροχής αδειών κατασκευής και οικοδόμησης διαφέρει ανάλογα με το project, ανάλογα με το έργο. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες υιοθετούν πολύ λογικά ε, πλαίσια, πολύ λογικούς κανονισμούς που δεν είναι υπερβολικά φορτωμένοι και αυστηροί και άλλες που δεν το κάνουν αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά ε, μια χώρα που ήρθε σε εμάς μερικές χώρες και είπε, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας είπε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κτηματολόγιο. Και εδώ βλέπουμε στην κατάταξή σας ότι δεν έχουμε καλή θέση, διότι ναι βεβαίως το κτηματολόγιό μας είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό, πολύ φορτωμένοι οι κανονισμοί, αλλά είναι πάρα πολύ σίγουρο, δεδομένου ότι άμα μπει στο κτηματολόγιο και λοιπά, μετά δεν γίνονται προσφυγές στα δικαστήρια, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι εμείς ε, πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα καθεστώς όπου το καλύτερο κτηματολόγιο θα επιτευχθεί όταν και ο αγοραστής και ο πολιτής ε, δώσουν τα χέρια και είναι ευχαριστημένοι και οι δύο. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία, το Ερμένο Βασίλειο, η Ελβετία που έχουν ένα πάρα πολύ ε, πιο εύκολο καθεστώς καταχώρησης ε, της, των αγοραπολισιών, δηλαδή ένα κτηματολόγιο ουσιαστικά, ε, και άλλες χώρες που έχουν ένα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία βάση στο επιχείρημα ότι εμείς ε, υποστηρίζουμε χώρες οι οποίες δεν έχουν ένα σωστό καθεστώς ε, καταχώρησης αγοραπολισιών ή και ότι με τον τρόπο αυτό διακυβεύουμε την ασφάλεια του συστήματος. Απλώς ε, τα, η συγκεκριμένη χώρα που ήταν χαμηλά στην κατάταξη είχε ένα πολύ φορτωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτό το κτηματολόγιο το οποίο ήταν και πολύ ακριβό. Γι' αυτό ήταν χαμηλά στην κατάταξη. Ε, γι' αυτό ακριβώς δίνουμε ανώτερη θέση στην κατάταξη σε χώρες οι οποίες συνδυάζουν μια πιο λογική και εύχρηστη λύση. Ό,τι αφορά τα θέματα διαφθοράς και το έβαλε σχετικό πίνακα, όπως ε, ανέφερε προηγουμένως η κυρία μας Καρντίνη που ανέφερε το θέμα της ε, διαφθοράς. Στο θέμα της ε, διαφθοράς υπάρχει ο, στον κατακόρυφο άξονα τον δείκτη αντίληψης περί διαφθοράς και, και στον άξονα των Χ η ταξινόμηση των των χωρών. Θα δούμε ότι αυτέ οι χώρες που έχουν χαμηλό επίπεδο επιχειρήν έχουν υψηλό επίπεδο διαφοράς και το αντίστροφο. Εάν πριν από 15 χρόνια η Παγκόσμια Τράπεζα είχε αναρωτηθεί τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μεταφέρουμε την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή κοινότητα σε ένα περιβάλλον λιγότερο διαφανές και λιγότερο διεθερμένο, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τίποτα πιο αποτελεσματικό από τη δημιουργία αυτών των δικτών εδώ πέρα ενισχύοντας και εισάγοντας ε, κίνητρα για την μείωση της υπερβολικού κανονιστικού πλαισίου των ε, πηγών διαφόρων προσκομμάτων, βλέπουμε ότι καθώς βελτιώνεται η ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς αυτές οι διαδικασίες δηλαδή γίνονται λιγότερο δαπανηρές και χρονοβόρες, μειώνονται και οι ευκαιρίες για διαφθορά και χρηματισμό. Και αυτό είναι εξαιρετικά ε, ενθαρρυντικό ως ε, απότοκο των ευρημάτων της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζουμε και του χρόνου να επαναλάβετε την άσκηση αυτή και να μας κάνετε αντίστοιχη παρουσίαση. Με μεγάλη με ευχαρίστηση θα επανέλθω, λέει ο Διευθυντής. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, πέρας της, ε, της ε, συνάντησης σήμερα, το επόμενο θέμα θα εξεταστεί και κλεισμένο των θυρών. Ζητώ λοιπόν από όσους δεν έχουν δικαιοδοσία να καταλήψουν την αίθουσα.